the most way I can Please, can you, can you please take your seats? We have to start a meeting. Για καθίστε παρακαλώ να αρχίσουμε. Okay. Allora, si è appena conclusa la riunione dei coordinatori. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνεδρία των συντονιστών, οι οποίοι αποφάσισαν να δεχθούν το αίτημα της κυρίας Βέρτμαν για να χαρακτηριστεί κατεπίγουσα η διαδικασία σχετικά με τις αναφορές που αφορούν τις απαγωγές ε, ανηλίκων στην Δανία. Απερίφθη αντιθέτως το αίτημα της κυρίας Διώτοβα να τοποποιηθεί η σύσταση σχετικά με τη 255 του 2013. Απερίφθη επίσης και το αίτημα Φερνάντες για την τροποποίηση της σύστασης για την 708 του 2013 και έγινε δεκτό το αίτημα του ιδίου συναδέλφου για την τροποποίηση της σύστησης για την 709 του 2013 διατηρώντας την συγκεκριμένη δηλαδή ε, αναφορά ανοιχτή. Έγινε δεκτό επίσης και το αίτημα των πρασίνων για την τροποποίηση της σύστασης για την F709-1 και την 694 του 13 οι οποίες παραμένουν ανοιχτές για την ημερήσια διάταξη δεν καταλήξαμε σε απόφαση γιατί δεν έχει ακόμα διανεμηθεί. Τώρα πλέον διανεμήθηκε η ημερήσια διάταξη και η τελική απόφαση για τις προτάσεις τις οποίες κάνει η Προεδρία θα τις έχετε στη διάθεσή σας αύριο το απόγευμα. Μέχρι αύριο το απόγευμα. Αποφασίστηκε παράλληλα σχετικά με την πρωτοβουλία των πολιτών να τροποποιηθούν οι οργανωτικές ε, ε, προεργασίες για την οργάνωση της πρώτης δημόσιας ακρόασης. Υπήρξε μια πρώτη ενημέρωση από πλευράς μου προς τους συντονιστές για την ε, αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος μέσω του καθορισμού κάποιων έκτακτων συνεδριάσεων της Επιτροπής μας που θα έχουν σαν στόχο την οργάνωση των πρωτοβουλειών αυτών Τέλος, σχετικά με το πόρταλ στο διαδίκτυο ε, υπήρξε αναβολή της δοκιμαστικής περίοδου. Θα ξεκινήσει στα μέσα Ιανουαρίου η δοκιμαστική λειτουργία και ε, έτσι ε, καθυστερεί για μια αντίστοιχη περίοδο η κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας. Πάντως εν τω μεταξύ θα οργανώσουμε μία συνεδρίαση ενημερωτική για τα μέλη της Επιτροπής για να μπορέσουν όλοι να κατανοήσουν το νέο μηχανισμό. Η θύρα αυτή δικτυακή δεν θα τεθεί σε λειτουργία αν δεν γίνει αντικείμενο έγκρισης από το σύνολο της Επιτροπής. Οι συντονιστές αποφάσισαν επίσης να εμείνουν στο θέμα της διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών γύρω από το θέμα του μη αποδεκτού της αίτησή μας για ειδική έκθεση για το Frontex, κάτι το οποίο είχε ζητηθεί από τον νέο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή η ε, διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών απέριψε όλες τέτοιου είδους εκθέσεις πρωτοβουλίες επειδή φτάνουμε υποτίθεται στο τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Αντίθετα εμείς ζητάμε να εμείνουμε στο αίτημά μας θεωρώντας ότι το θέμα του Frontex είναι κατεπήγον και θα αποστείλουμε ένα αίτημα εκ νέου. Ταυτόχρονα έχει αποφασιστεί η ένταξη στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών μας τον μήνα Φεβρουάριο και τον μήνα Μάρτιο κάποιων θεμάτων αρκετά ευαίσθητων. Δηλαδή, τον Φεβρουάριο θα συζητηθούν οι αναφορές για τις απαγωγές ανηλίκων στην Δανία και επίσης η κατάθεση της προκαταρκτικής έρευνας για τα θέματα της εφαρμογής της διαδικασίας της πρωτοβουλίας των πολιτών και τον Μάρτιο θα ασχοληθούμε με τις αναφορές που αφορούν πάντα α, α, τέτοιες απαγωγές στην Αυστρία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω σχετικά με τη συνεδρίαση των συντονιστών. Περνώ στο επόμενο θέμα πλέον της ημερήσιας διατάξεως, δηλαδή την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. έχουμε σαν πιο σημαντικά σημεία οκτώ αναφορές σχετικές με τα της μετανάστευσης, τα δικαιώματα των προσφύγων και τις διαδικασίες γύρω από το δικαίωμα χορήγησης ασύλου. Έχουμε επίσης ε, και το θέμα της μονάδας ε, παραγωγής αερίου στο Ρωμανβίλ στη Γαλλία Έχουμε την ψηφοφορία για την αποστολή στην Γαλλικία. Τώρα πάντα για την ημερήσια διάταξη έχουμε λάβει σαν Προεδρείο ένα αίτημα τροποποίησης για το σημείο 14 αίτημα Μπέκερ το οποίο συνοδεύτηκε επίσης και από τον πρώτο υπογράφοντα την αναφορά, γιατί δεν μπορούν να είναι παρόντες ε, οι αναφέροντες και αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση. Έχει ζητηθεί επίσης ε, και η αναβολή από πλευράς των συναδέλφων Γιάρε και Μποστινάρου ε, του σημείου 16 περιβάλλον σχετικά με την υπόθεση της Ρώσια Μοντάνα. Ε, θεωρήθηκε χρήσιμο από πλευρά των δύο συναδέλφων και τεκμηρίωσαν ε, τα επιχειρήματά τους προς όφελος, αν θέλετε, της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του αναφέροντος ε, να υπάρξει μια κάποια αναβολή για λίγες εβδομάδες. Βέβαια, το αίτημα αυτό έφτασε αρκετά καθυστερημένα και δεν μπορέσαμε εκ των προτέρων να οργανώσουμε τα της μετακίνησης του αναφέροντος, ο οποίος είναι εδώ ανάμεσά μας. Οπότε το αίτημα του κυρίου Μποστουνάρου και του κυρίου Γιάρη δεν μπορούμε να το κάνουμε δεκτό. Σχετικά τώρα με την ομάδα αναφορών, την σχετική μετά της μετανάστευσης, έχουμε παρόντες παρούσα μάλλον την κυρία Καλάιτενεν ε, που είναι εκπρόσωπος της ε, Frontex και θα της δώσουμε το λόγο όταν ασχοληθούμε με τις σχετικές αναφορές. Να προσθέσω επίσης, δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, κάποια μέλη επίσης εδώ παρόντα ε, ότι ενημερώσαμε τα θέματα αυτά και, και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ γιατί είναι και δική της αρμοδιότητα. Έχουμε και το σημείο 15, ο αναφέρον δεν μπορεί να είναι παρόν και έχει ε, διανεμηθεί ένα σημείωμα εκ μέρους του σχετικά με την ψηφοφορία για την Γαλλικία ορίστηκε η ψηφοφορία να ξεκινήσει τη 18η απογευματινή μετά από αίτημα του κυρίου Μπουλάν και δεν έχουν υπάρξει άλλες αιτήσει τροποποίησης της ημερησίας διατάξεως την οποία πλέον σας καλώ να δεχτείτε. Η κυρία Άουκεν έχει τον λόγο μετά ο κύριος Μποστινάρου. Θα μιλήσω την δανική. Κοιτάξτε, ε, στην Επιτροπή μας Όσοι συνηθίζετε θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα και αλλού που ανυπομονούν τόσο πολύ να γνωρίζουν πώς αντιδρά, πόσο γρήγορα αντιδρά η Επιτροπή μας σε ορισμένες αναφορές. Δεν θα ήταν αποδεκτό να κάνουμε τίποτε διαφορετικό. Μετά. Για το άλλο θέμα, το άλλο. Α, όχι, ας μέρα μείνω σε αυτό. Αφήνω το άλλο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θέλω να κάνω μερικές αποσαφηνήσεις. Δεν θα σχολιάσω εδώ μέσα μια συζήτηση που κάναμε στους συντονιστές, αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω πώς έφτασε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για μέθοδο που μου θέτει πολλά ερωτήματα. Εδώ δεν αφισβητώ ούτε τη δραστηριότητα των συντονιστών ούτε της γραμματείας. Αλλά την πρόταση αυτή της συναδέλφου Χάουκεν για την εκμετάλλευση των χρυσορυχίων στη Ρουμανία την είχαμε ξανασυζητήσει. Πρώτον, η Βουλή της Ρουμανίας δεν θέλησε δύο φορές απέσυρε ένα τέτοιο αίτημα και αρνήθηκε ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και την περασμένη Τρίτη πήραμε απόφαση πολύ καινοτόμα θα έλεγα, στη Ρουμανία εννοώ την Τρίτη, καινοτόμα απόφαση σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές. Εδώ και δύο χρόνια μας είπε η Κομισιόν κάτι που το επανέλαβε με τα ίδια λόγια τον Νοέμβριο. Δεν έγινε καμία μελέτη αξιολόγηση για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και γι' αυτό δεν μπορεί να αποφανθεί, είπε. Τι μπορούμε να προσφέρουμε σήμερα για τον αναφέροντα τον οποίο χαιρετίζω εδώ. Μπορούμε να του προτείνουμε να κλείσουμε την αναφορά. Εγώ είμαι κατά. Θέλω να παραμείνει ανοιχτή. Τι μπορούμε να του προτείνουμε λοιπόν. Να γίνει συζήτηση χωρίς κανένα επιχείρημα ούτε υπέρ ούτε κατά και τι να πούμε στην Κομισιόν, τίποτα επίσης. Διότι προς στιγμήν το πρόγραμμα αυτό, το σχέδιο αυτό, τα χρυσορυχεία δηλαδή, βρίσκεται σε άλλη φάση από εκείνη πριν δύο χρόνια όποτε έγινε η πρώτη συζήτηση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να την ξανασυζητήσουμε άλλη φορά όταν θα έχουμε άλλα στοιχεία. Κοιτάξτε, περί αυτού πρόκειται, θα ξεκινήσω από το τέλος. Πρόκειται για το σημείο υπερθμών 16. Ο κ. Μοντάνα και εγώ θέλουμε να κρατήσουμε ανοιχτή την ε, ε, αναφορά και προ όφελο της διαδικασίας ε, και του αναφέροντος. Λυπηρό είναι αυτό, αλλά εγώ διατηρώ το δικαίωμά μου, θέλω να ψηφίσουμε και θέλω το 16 να φύγει από την ημερήσια διάταξη. Διότι η δική μου η ομάδα ποτέ δεν συμφώνησε να εξεταστεί σήμερα το θέμα αυτό και αυτό είναι και προ όφελο ε, των αναφερόντων. Ε, Παναλαμβάνω λοιπόν για άλλη μια φορά η δική μου πολιτική ομάδα, το ΕΛΚ, θέλει να κρατήσει ανοιχτή αυτή την αναφορά και να τη βγάλει από την ημερήσια διάταξη. Εδώ ζητιέται λοιπόν ψηφοφορία. Την Επιτροπή μας λοιπόν την παρουσιάζουμε σαν επιτροπή που δεν έχει κανόνες σταθερούς. Κάνει ανάλογα με την περίπτωση. Ενώ εδώ εκπροσωπούμε τους πολίτες, καλέσαμε τον αναφέρον, τους αναφέροντες. Η αναφορά έχει πολύ καιρό που υποβλήθηκε, που πρώτο υποβλήθηκε. Και αν ο κύριοι Γιάρ στην Άρου κάνουν το δικό τους, αν περάσει το δικό τους, δεν ξέρω τι θα απογίνουμε. Πολλές φορές παραμένουν εκκρεμούσες αναφορές και σε άλλα κοινοβούλια. Οι πολίτες μας προσέχουν στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ουγγαρία. Όλοι προσέχουν να δουν πώς θα χειριστεί η Επιτροπή Αναφορών αυτό το θέμα των χρυσορυχίων. Εάν λοιπόν δεν πούμε τίποτα ρητό, ούτε η Κομισιόν πει τίποτα, δεν είναι θετικό αυτό για μας. Να φαίνεται δηλαδή ότι για ένα θέμα όπου υπάρχουν διαμάχες δεν κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό παρακαλώ να παραμείνει η διάταξη ως έχει. Και να χειριστούμε, να διεκπαιρεώσουμε την αναφορά όπως προβλεπόταν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστώ μερικά δευτερόλεπτα μόνο. Δεν χρειάζεται να αρχίσει εδώ ολόκληρη συζήτηση. Έχουμε την πρόταση Χάουκεν και έχω και εγώ μια πρόταση εξ ονόματος της ομάδας μου. Να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε. Έχουμε εδώ τους συναδέλφους βουλευτάς. Να ψηφίσουμε. Για το τι θα γίνει με την αναφορά αυτή. Τελεία και παύλα. Και μετά θα ακολουθηθεί η μερίσια διάταξη ως είχε. Αυτό είναι νομίζω το λογικότερο. Υπάρχουν λοιπόν δύο προτάσεις να ψηφίσουμε. Να σας εξηγήσω την αντιπρόταση. γιατί ίσως έτσι να δούμε τα πράγματα σαφέστερα. Έχουμε μπροστά μας, μεταξύ μας, τον αναφέροντα. Εγώ είχα δεχτεί την πρόταση της Προέδρου, αλλά ας προσπαθήσουμε να συνοηθούμε για το 16 να ακούσουμε τουλάχιστον τον αναφέροντα για να είμαστε πιο πληροφορημένοι και μετά να περάσουμε στο επόμενο σημείο και να ακούσουμε την Κομισιόν. Αλλά ας αφήσουμε τον αναφέροντα να μας πει αυτά που θέλει. Αφού ήρθε, να μην του κλείσουμε την πόρτα στα μούτρα. Ένα μόνο λεπτό όμως κύριε Μποστινάρου, ε. Μα δουλεύει το μικρόφωνο μου, γιατί μου λέτε ότι δεν δουλεύει. Λοιπόν, κανείς δεν αφισβητεί τα δικαιώματα του αναφέροντος. Δεύτερον, εγώ δεν χρειάζομαι μαθήματα να μου δίνετε μαθήματα ή να μου δίνουν μερικοί συνάδελφοι. Και τρίτον, ποτέ δεν θα δεχτώ να κατηγορείται η χώρα μου όταν δεν εξυπηρετεί αυτό τα συμφέροντα κανενός αναφέροντα. Αυτό δεν το λέω για να αυξηθώ το γόητρό μου στη Ρουμανία. Κάνω ό,τι μπορώ για να εξυπηρετήσω όσο το δυνατόν καλύτερα τα συμφέροντα των αναφερόντων όταν υπάρχουν επιχειρήματα. Και τέλος, ούτε εγώ ούτε ο Πίτερ δεν καλέσαμε τον αναφέροντα, αλλά άλλοι. So, to clarify ναι. Καλά, για να τα ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Πρέπει να ψηφίσουμε κυρία Χάουκιν διότι το θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη και κάθε φορά ψηφίζουμε την έγκρισή της. Είμαστε ήδη στο δεύτερο σημείο που είναι η έγκρισή της. Τι άλλο να σας κάνω. θα ψηφίσουν οι συνάδελφοι, τα πλήρη μέλη μόνο. Και προσθέτω κάτι ιδιαίτερα για τον κύριο Μποστινάρο και τον κύριο Γιάρ που είπαν ότι δεν ήταν σωστό διαδικαστικά αυτό που έγινε. Σας υπενθυμίζω ότι το αίτημα της κυρίας Χάουκεν είχε προωθηθεί στις 28 Νοεμβρίου πρώτη φορά και μοιράστηκε σε όλους τους συντονιστές. Όλοι οι συντονιστές το δέχτηκαν στις 29 και όλα αυτά είναι γραπτά, κύριε Γιάρο. Τα έχω εδώ, έχω έγγραφα και σας θα εξηγώ. Μετά, η ημερήσια διάταξη 3 Δεκεμβρίου διανεμήθηκε και στις 5 Δεκεμβρίου η ημερήσια διάταξη που ημεριαλάμβανε και αυτό το θέμα εγκρίθηκε πάλι από τους συντονιστές. Μετά ζητήθηκε η αλλαγή και είπα γράψτε μου και επιχειρήματα για το αίτημα αυτό της αλλαγής και πέστε μου ποιος υποστηρίζει από τους συντονιστές μας το αίτημα της αλλαγής. Στις, 12, στις 11 Δεκεμβρίου έλαβα και άλλο αίτημα του κυρίου Γιάρ, εκτός από του κυρίου Μποστινάρου, για αλλαγή της ημερήσιας διάταξης. Και προσπάθησα μέσω της γραμματείας να αλλάξω την ημερήσια διάταξη σητώντας, ρωτώντας τον αναφερόμενο αν ήταν δυνατόν να αλλάξει αυτά που είχε προβλέψει επειδή όμως είδαμε ότι δεν μπορούσε ο αναφερόμενος ήρθε, είναι εδώ μεταξύ μας και είπα να του, είπα να του δώσουμε το λόγο, ούτως ή άλλως. Αυτά είναι τα διαδικαστικά λοιπόν και δεν μπορώ να αποφύγω την ψηφοφορία για την ημερήσια διάταξη. Διότι αυτή, αυτός είναι ο κανονισμός μας. Πρέπει να ψηφίσουμε την, την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. για διάφορα τμήματα, σε διάφορα τμήματα, γιατί το μόνο θέμα, αν δεν απατώ με το μόνο θέμα όπου διαφωνείτε είναι αυτό, το 16. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι εγκρίνεται η μυρίσια διάταξη εκτός από το 6 λέει τώρα η ομιλήτρια όπου θα ψηφίσουμε χωριστά. Ποιος είναι λοιπόν υπέρ της διατήρησης του 16 αυτή τη φορά στην σημερινή ημερήσια διάταξη. Υπέρ, υπέρ της διατήρησης. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, έξι. Ποιος είναι κατά. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά. Εγώ Υπέρ, υπέρ, υπέρ. Εγώ μέτρησα 7, αλλά θα ξαναμετρήσουμε. Ξανά. Κατά, ξανά. Κατά. Α, 6, 6. 6, 6. 6, 6. παραμένει στην ημερήσια διάταξη. Παραμένει. Has been approved as said. Uh, as far as the item 3 is... Τώρα για το 3, όπως πάντα είχαμε μοιράσει έναν κατάλογο νέων αναφορών με τη προτινόμενη κρίση μας δεν έλαβα σχόλια μέχρι να τελειώσει η συνεδρίαση θα εγκριθεί ο κατάλογος αυτός ως είχε δεν έχω άλλες ανακοινώσεις το 4 όχι Μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στο 6. Έχουμε 8 αναφορές που υποβλήθηκαν από τη Λούση Χάρντ και άλλους. Ελίζαμπετ Σμόκ και άλλους. Μπέρναρντ Σέγγεν Ρενάτο Λέλη που εκπροσωπούν που εκπροσωπεί μια Ιταλική οργάνωση άλλοι προασμούντες, Φάισερα, αρμαϊσμούντες και Φάισερα και τα Μια άλλη από την τώρα Τεματία, Τσέζαρε Ρίτσι, και η τελευταία από τον Εμιλιάνο Φρατέλο. Για όλες αυτές τις αναφορές παρίσταται σήμερα μόνον ο κύριος Εμιλιάνος Φρατέλο στον οποίο και δίνω το λόγο για πέντε ολόκληρα λεπτά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την πρόεδρο της Επιτροπής και τους ε, βουλευτές ε, και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας έδωσαν τη δυνατότητα να έρθουμε σήμερα εδώ για να εκπροσωπήσουμε τη δική μας την άποψη για ένα θέμα που είναι τόσο σημαντικό. Έχει και ηθική σημασία και βαρύνουσα σημασία. Πέντε λεπτά μου έχετε δώσει. Σημαίνει κάτι, λέει Πρόεδρος. Ήρθαμε λοιπόν εδώ για να μιλήσουμε για τη μετανάστευση και για τα διάφορα θέματα που αποτελούν το φαινόμενο αυτό. Η δική μας η χώρα, κυρίως η Ιταλία, στην Λαμπεντούζα, βιώνει ε, την τραγωδία όλων αυτών των ανθρώπων που προσπαθούν ε, να έρθουν στην Επιρώμα. μας. Υπάρχει λοιπόν αυτό το δράμα της Λαμπεντούζα και από εκεί ορμόμενοι σκεφτήκαμε να κινητοποιηθούμε και να γνωστοποιήσουμε στην κοινή γνώμη ένα θέμα το οποίο είναι περισσότερο πολιτιστικό. Πριν λοιπόν φτάσουμε στο θέμα της αναφοράς, θελήσαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών, όλων εκείνων που ζουν το πρόβλημα ε, επειδή δέχονται τις, ε, τους πρόσφυγες και ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να μας κατευθύνουν στη σωστή πολιτική τοποθέτηση. Στην Ευρώπη λοιπόν η μετανάστευση είναι η προσέγγιση ενός πολύ συγκεκριμένου προβλήματος από το 1988 στα σύνορα της Ευρώπης έχουν πεθάνει περίπου 19.000 άνθρωποι, εκ των οποίων 2.000 περίπου μόνο το 2011. 550 ε, ε, την επόμενη χρονιά και εξίσου ε, σημαντικός αριθμός το 2013. Όλα αυτά βασίζονται σε στοιχεία που υπάρχουν στον διεθνή τύπο τα τελευταία 7 χρόνια. Και αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι κανείς δεν ξέρει ακριβώς πόσοι πνίγησαν, από αυτούς δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Ε, οι, γονείς, οι οικογένειές τους εδώ και χρόνια διερωτώνται τι ακριβώς συνέβη με τα παιδιά τους που έφυγαν για την Ευρώπη και δεν γύρισαν ποτέ. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα και θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει μια άμεση οργάνωση που να αφορά στην ε, υποδοχή των προσφύγων. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να παρεύουμε σε θέματα ελέγχου και ασφάλειας των ευρωπαϊκών συνόρων. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διασφάλιση της ζωής των ανθρώπων αυτών και θέλουμε όλα αυτά να τα κάνουμε με έναν τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμός για τη μετανάστευση, να μπορούμε να συνεργαστούμε. Οι ευρωπαϊκές χώρες πλήττονται από ε, ροές μετανάστευσης, ε, υπάρχουν χώρες προέλευσης των μεταναστών, χώρες τράνζιτ, διαμετακόμιση σε χώρες υποδοχής και οι πολίτες λοιπόν έχουν να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις ε, θεσμικές αποφάσεις. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια υποδομή που θα επιτρέπει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να ζουν ε, όπως ε, πρέπει, όπως προβλέπετε, το 2014 είναι καθοριστική χρονιά η Ελλάδα και η Ιταλία που δέχονται πολλές μεταναστευτικές ροές θα αναλάβουν την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα λοιπόν σε δύο εξάμεινα μπορούν οι χώρες αυτές ε, να εξετάσουν γενικότερα την κατάσταση στη Μεσαίγειο όσον αφορά τις ροές μετανάστευσης, έτσι ώστε να υπάρχει και μία μόνιμη πλατφόρμα αντιμετώπισης του προβλήματος. Ζητάμε λοιπόν από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δική μας την πρόταση, να υπάρχει δηλαδή πολυεπίπεδη συνεργασία σταθερή όχι μόνο ανάμεσα σε κράτη αλλά ανάμεσα και σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, σε πανεπιστήμια, σε διάφορους θεσμούς. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να ανταποκριθεί. Η συνεργασία λοιπόν πρέπει να είναι θεσμική και αυτή που υπήρξε έχει ήδη καταδείξει ότι μπορεί να υπάρξει κάποια ταύτιση απόψεων. Μέχρι τώρα η σκληρή στάση δεν έχει λειτουργήσει. Ναι. Οφείλουμε λοιπόν να καταφύγουμε στη διπλωματία η οποία ξεκινάει από γενικά αρχές και φτάνει στις μεταναστευτικές ροές. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να χειριστούμε το φαινόμενο αυτό ε, και κατά τα άλλα νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ε, την δυνατότητα έπαρξης ενός μόνιμου συμβουλίου για τη μετανάστευση. Ε, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να συνεργαστούν. Όλα αυτά θα επιτρέψουν στην κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης να μην δέχονται αγόγγιστα τις αποφάσεις και τις επιλογές των πολιτών, αλλά να συμμετέχουν και οι ίδιες στην κατάρτιση επιλογών, κυρίως για, τους, για τις χώρες πρώτης υποδοχής. Ε, δεν ε, πρέπει να καταλήγουμε στις κλασικές αποφάσεις, αλλά να δημιουργήσουμε τέτοια υποδομή που θα επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να περιορίσουμε και τους παράνομους μετανάστες. Ο εθελοντισμός και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, είναι εκείνες που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υποδοχή των μεταναστών. Δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένας μηχανισμός που θα τους καθιστά πρωταγωνιστές, κυρίως στη φάση κατά την οποία χαράσσονται οι μεταναστευτικές πολιτικές. Το ίδιο και για τον Νότο ε, μια κοινωνία των πολιτών ε, υπάρχει σε πολλές χώρες ε, του Μαγκρέπ, κυρίως στην Αίγυπτο. Αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη υποδοχή των μεταναστών, καλύτερη οργάνωση των ροών Κατόπιν τούτου, τελειώγοντας, θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία των πολιτών. Και θεωρώ επίση ότι αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δώσουμε ένα πολιτιστικό παράδειγμα ε, για, τις, για τη μετανάστευση. Ε, είναι λοιπόν σημαντικό να ε, μην υπάρχει ξενοφοβία και να υπάρχει ένας πραγματικός πολιτισμός υποδοχή στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντιμπλάζη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τους αναφέροντες μετά το ναυάγιο της Λαμπεντούζα. Την επομένη του τραγικού συμβάντος τον προηγούμενο Οκτώβριο ξεκίνησε τη διαδικασία για να βρει νέες δράσεις στον τομέα της μετανάστευσης που θα ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις των Ευρωπαίων πολιτών και των ηγετών έτσι ώστε να σταματήσουν φαινόμενα σαν αυτό της Λαμπεντούζα. Επισκέφθηκε στις 9 Οκτωβρίου ο κύριος Μπαρόζο τη Λαμπεντούζα, ξεκίνησαν αμέσως συγκεκριμένες δράσεις για να απαντήσουμε στην πρόκληση. Το Frontex ενίσχυσε την παρουσία του και ε, δόθηκαν πιστώσεις και στην Ιταλία και σε άλλες μεσογειακές χώρες για να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα μεταναστευτικά ρεύματα. Παράλληλα, μετά από αίτημα των Ιταλικών Αρχών και του Συμβουλίου, δημιούργησε μία task force για την Μεσόγειο. Εντόπισε οκτώ δράσεις για να αντιμετωπίζει καταστάσεις όπων της Λαπεντούζα και ήρθε σε επαφή και με άλλους εμπλεκομένους όπως επίσης την ύπατη αρμοστία για να οργανωθούν οι δράσεις αυτές με συμμετοχικό τρόπο και όχι σαν κάτι το οποίο αποκλειστικά οργανώνεται από τα ίδια τα κράτη. Αυτά περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε δεκτή στις 4 Δεκεμβρίου. Συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Νομικών Υποθέσεων στις 5 Δεκεμβρίου και είναι τώρα στην φάση αποστολής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ανακοίνωση αυτή προσπαθεί να απαντήσει στις βασικές αιτίες ε, και τα λειτουργικά προβλήματα της περίπτωσης Λαμπεντούζα. Αυτό δεν αρκεί βέβαια, απαιτείται εμπλοκή μακροπρόθεσμη και γι' αυτό ζητάμε από τους αναφέροντες να απαντήσουν και να πάρουν μέρος στην παρούσα διαβούλευση που έχει ξεκινήσει ε, στην Γενική Διεύθυνση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον της πολιτικής μας δράσεις βραχυπρόθεσμες έχουν ήδη αποφασιστεί, αλλά πρέπει να γίνουν και διάφορα περισσότερα πράγματα μακροπρόθεσμα στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας, της κοινωνίας των πολιτών και μετά από την υιοθέτηση του κοινού συστήματος από πλευράς του Συμβουλίου και μέσω νέων νομοθετικών μέτρων. Ε, όπως μας υπενθύμησαν ε, οι αναφέροντες, το μέλλον ε, στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων είναι υπό επεξεργασία στην παρούσα φάση και γι' αυτό θα πρέπει όλοι να τηρήσουμε στάση αναμονή σε μια πρώτη φάση αυτό. Βέβαια καλύπτει παρόλα αυτά αρκετές από τις αναφορές που κατατέθηκαν σήμερα. Θα είμαι στη διάθεσή σας για τα ειδικότερα θέματα από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος, ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex μάλλον έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Αναφορών που με προσεκάλεσε και μου έδωσε τη δυνατότητα να διευκρινίσω κάποιες πλευρές της δράσης μας οι οποίες σχετίζονται ε, με ε, την φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Όπως ε, είπε ήδη ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή είναι βασική προτεραιότητα στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων, όχι μόνο από την 3η Οκτωβρίου και μετά, αλλά και πριν. Η δουλειά της Task Force Μεσόγειος αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται και το Frontex συμμετέχει ε, στις εργασίες αυτής της Task Force. Να πω τώρα κάποια γενικά για το ποιες είναι οι τάσεις τις οποίες βλέπουμε εμείς στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς δεν έχω να σας δώσω νέα καλά η κατάσταση στην κεντρική Μεσόγειο, στην κεντρική Μεσόγειο επαναλαμβάνω, είναι πολύ σοβαρή και αντίθετα από τον προηγούμενο χρόνο, στην παρούσα φάση τα μεταναστευτικά ρεύματα αυξάνονται. Κανονικά κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου έπρεπε να μειούνται, αλλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο φέτος. Το άλλο είναι ότι ήδη είδαμε ότι τα πλεούμενα τα οποία προσφέρουν οι διαμεσολαβητές τους παράνομους μετανάστες είναι όλο και πιο ανασφαλή, βυθίζονται όλο και περισσότερα και στερούνται γενικά κάθε συνθήκης για αξιοπρεπή μεταφορά. Δεν έχουμε και στον τομέα αυτό να μεταφέρουμε κάτι το καλό δηλαδή. Ταυτόχρονα αν δούμε τη γεωπολιτική κατάσταση και ελέγξουμε τις βασικές αιτίες, θα δούμε ότι υπάρχει ένα υψηλότατο επίπεδο αβεβαιότητας στην περιοχή. Τρεις είναι οι βασικές χώρες από τις οποίες προέρχονται οι παράνομοι μετανάστες, Συρία, Ερυθρέα και Σομαλία και ακολουθούνται από ε, πολίτες του Αφγανιστάν. Νομίζω ότι τα ονόματα αυτών των χωρών σας δείχνουν γιατί ασχολούμεθα με αυτό το φαινόμενο. Έχουμε δύο πολύ σοβαρά θέματα ε, γεωγραφικά. Το κέντρο της Μεσογείου καταρχάς που συνδέουν την Ιταλία όχι μόνο με την Λιβύη αλλά και με την Αίγυπτο από κοινού. Πρόκειται για δύο ροές ουσιαστικά οι οποίες έχουν σαν στόχο την Ιταλία. Αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι η αριθμή και η πίεση στην παρούσα φάση εξαρτάται από την συγκυρία. Αλλά παρόλα αυτά μιλάμε για περισσότερο κόσμο από ότι το 2011 κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης. Ένα άλλο θέμα που αφορά τα επίγεια σύνορα είναι τα σύνορα κυρίως Τουρκίας-Βουλγαρίας. Η αύξηση των ε, εισόδων παρανόμων μεταναστών είναι χωρίς προηγούμενο και οι Σύριοι είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούν το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο ποσοστό. Η Task Force για τη Μεσόγειο λοιπόν είπαμε ότι προτείνει συγκεκριμένες δράσεις που καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες. Υπάρχουν και κάποια θέματα που άπτονται των εξωτερικών υποθέσεων, της ενίσχυσης των νομικών διαδικασιών, της καταπολέμησης εγκληματικών οργανώσεων και επίσης και κάποιες επιτόπου λειτουργίες και δράσεις με βάση το Frontex. Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι είναι δραστηριότητες οι οποίες ξεκινούν από τις δράσεις των ιδίων των κρατών μελών. Οι τοπικές αυτές δράσεις συμπληρώνονται από περιφερειακές συνεργασίες ανάμεσα στις διαφορετικές ε, χώρες στα πλαίσια του European Patrol Network. Από εκεί και πέρα έρχεται το Frontex και συντονίζει τις δράσεις περισσότερων χωρών. Και υπάρχουν από εκεί και πέρα και κάποιες άλλες μεμονωμένες δράσεις κρατών μελών, όπως σαν παράδειγμα η επιχείρηση Mare Nostrum από την Ιταλία. Ε, όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία χρήζουν ε, υψηλού επίπεδου συντονισμού και δεν είναι εύκολο να το πετύχουμε αυτό. Παράλληλα θα πρέπει εμείς να έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη για το τι συμβαίνει. Η βασική πρόκληση είναι να είμαστε ικανοί, να εντοπίζουμε, να ανοιχνεύουμε μικρά πλεούμενα και αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα στην παρούσα φάση. Αυτή είναι η αδυναμία μας σε σχέση με τις επιχειρησιακές μας ικανότητες. Τώρα, για το Frontex και το ρόλο του. Το Frontex λειτουργεί συντονιστικά. Εμείς συντονίζουμε τις επιχειρησιακές δράσεις των κρατών μελών. Όλες οι κοινέ επιχειρήσεις ελέγχονται από το κράτος μέλος κάθε φορά στο οποίο το έδαφος διεξάγεται η επιχείρηση. Ποια είναι η πρόκληση την οποία έχουμε μπροστά μας. Ποια η δυσκολία είδαμε κάποιες μειώσεις των πιέσεων σε σχέση με την βούληση των κρατών μελών να θέσουν στη διάθεση του Frontex τους εμπειρογνώμονες και τα τεχνικά μέσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται στην παρούσα φάση, μια λιγότερη προθυμία θα έλεγα. Ένα άλλο θέμα είναι το μέγεθος, η κλίμακα των επιχειρήσεων του Frontex. Εδώ τα μέσα ενημέρωσης δίνουν λανθασμένη εντύπωση. Τυπικά μία επιχείρηση όπως η Ιταλική Ερμές, Ερμής ή Ενίας, η συμμετοχή του Frontex είναι δύο αεροσκάφη και ένα σκάφος, ένα πλεούμενο. Αν τα συγκρίνουμε αυτά με τις ικανότητες που έχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ιταλία, μιλάμε για κάτι το πάρα πολύ μικρό. Είναι σαφές λοιπόν πρέπει να γνωρίζουμε την κλίμακα παρέμβασης. Ε, μας δώσαν στο τέλος του χρόνου 8 εκατομμύρια ε, επιπλέον ευρώ. Τα πήραμε με μεγάλη καθυστέρηση και καλούμεθα με τις πιστώσεις αυτές να διασφαλίσουμε τη συνέχεια των επιχειρήσεων στις πιο κρίσιμες περιοχές της Μεσογείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις εντατικοποιήσαμε τις επιχειρήσεις μας. Έχουμε επίσης προγραμματίσει ε, κατεπηγόντως για το 2014 και υπολογίσαμε ότι θα απαιτηθούν άλλα 14 εκατομμύρια για να διασφαλίσουμε τη συνέχιση των επιχειρήσεων και να διασφαλίσουμε επίσης και εντατική παρουσία μας σε ορισμένες από τις επιχειρήσεις. Αυτές είναι οι δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Μια τελική παρατήρηση μεθοριακός έλεγχος και θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι για μας προτεραιότητα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι προτεραιότητα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν, όχι μόνο να σεβόμεθα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά να προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια του σύγχρονου τρόπου διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δημιουργήσει ένα καλό προηγούμενο θα έλεγα. Πρώτον, σχεδιάζουμε σωστά τις δράσεις μας. Βλέπουμε ε, τι δομές χρησιμοποιούμε στις επιχειρήσεις αυτές. Δεύτερον, η σωστή κατάρτιση των συμμετεχόντων στις ε, έρευνες αυτές και στις προσπάθειες. Υπάρχει επιτόπου εκπαίδευση, ιδιαίτερα εκεί όπου συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Έχουμε και κάποιες άλλες οριζόντιες δραστηριότητες, όπως η κοινότητα των ε, μεθοριακών ε, φρουρών, σκοπών αν θέλετε, και κάποια άλλα μέσα αύξησης των ικανοτήτων ε, των κρατών μελών στον τομέα αυτό της φύλαξης των συνόρων πάντα τύχαμε τις στήριξης δύο καινοτομιών από πλευράς του νέου κανονισμού Frontex. Πρώτον, το φόρουμ διαβούλευσης και δεύτερον, η υπηρεσία ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και ε, τα, οι δύο αυτοί παράγοντες λειτουργήσαν θετικά στην προσπάθειά μας. Τελικά λοιπόν ανησυχούμε, είναι αλήθεια για την κατάσταση Πράγματι το Frontex όμως κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να παράσχει όλες τις δυνατότητες τις οποίες χρειάζεται ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συντονίζει σωστά τις προσπάθειες των κρατών μελών. Στα πλαίσια του ευρυτέρου πλαισίου του Task Force Μεσόγειος πάντα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Τώρα θα αρχίσει η συζήτηση. Πρώτος ο κύριος Μέγερ. Θέλω να ευχαριστήσω τον αναφέροντα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι είναι πολύ επίκαιρη συζήτηση αυτή, ένα θέμα τόσο ευαίσθητο, γιατί πάρα πολλοί είναι αυτοί που χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τραγωδία της Λαμπεντούσα νομίζω ότι είναι το βασικό σημείο μιας τραγωδίας που θα έλεγα κεντρικής και σε σχέση με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι είτε οικονομικοί μετανάστες, είτε ετούντες άσυλο ή που θέλουν να μπουν στη διαδικασία να ζητήσουν άσυλο. Είναι μια τραγωδία που συνεχίζει να εξελίσσεται. Νομίζω ότι η απόρριψη του Προέδρου Μπαρόσο στη Λαμπεντούσα αντικατοπτρίζει σωστά την κατάσταση η οποία επικρατεί και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το οξυμένο αυτό πρόβλημα. Δυστυχώς είμαστε μακράν του να σεβόμαστε το άρθρο 3 της, ε, α, της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να επιλέξει τον τόπο κατοικίας του. Είναι επίσης το άρθρο 13, συγγνώμη, αλλά είναι επίσης ότι δεν είμαστε σε θέση έτσι κι αλλιώς όπως είναι τα πράγματα τώρα να δώσουμε εγγυήσεις για την εφαρμογή της αρχής της χορήγησης ασύλου και του δικαιώματος που αντιστοιχεί σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν νομοθετεί ή όταν συνομοθετεί δίνει την αίσθηση ότι αντιμετωπίζει αυτούς που δεν έχουν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα σαν, παρα, σαν εγκληματίες, σαν παρανόμους μάλλον και έτσι δημιουργείται ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Νομίζω λοιπόν, και αυτή είναι μια προσωπική μου δεοντολογική άποψη, ότι αυτός που δεν έχει τα σωστά χαρτιά δεν είναι παράνομος. Εμείς ε, είχαμε ψηφίσει στην αρχή της κοινοβουλευτικής ε, περίοδου ε, την ε, οδηγία για την παλινόστηση την υποχρεωτική και ξέρουμε ότι δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα, κρατούνται οι άνθρωποι αυτοί ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έδειξε ένα καλό πρόσωπο και αυτά ακριβώς προκαλούν αυτό που είπα ήδη, την ξενοφοβία και τον λαϊκισμό. Δημιουργούνται νέα κινήματα ρατσιστικά, φασιστικά σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε όπως ε, είπα μακράν του να κάνουμε σεβαστές τις αρχές αυτές των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομίζω ότι όσο και να προσπαθεί να πιέσει κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να καταλήξει κάπου δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με ελάχιστα μέσα και δυστυχώς ο κόσμος συνεχίζει την προσπάθεια να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να χτίζει τύχη και ο κόσμος χάνει τη ζωή του προσπαθώντας να διασχίσει τα τείχη αυτά. Είδαμε τι γίνεται στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού ο κόσμος με τον ένα τρόπο ή τον άλλο θα συνεχίσει να προσπαθεί να έρχεται και θα μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χάνει και τη ζωή του, μετακινούνται ε, οικογένειες ε, για να ξεφύγουν από τη φρίκη του πολέμου, για να ξεφύγουν από την απάνθρωπη κατάσταση στην οποία έχουν στις χώρες προέλευσης. Είναι λοιπόν καιρός να αντιδράσει πλέον η κοινωνία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προκαλέσει μια αλλαγή νοοτροπιών, στάσεις και να πάρουμε νομοθετικά μέτρα έτσι ώστε κάποια στιγμή το 2013 να γίνει πραγματικότητα στα πλαίσια μιας ανθρωπιστικής στάσης σεβασμού αυτών που απειλείται η ζωή τους. Ο κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για τη συζήτηση που γίνεται σήμερα. Είναι πραγματικά ένα ε, πάρα πολύ σημαντικό και επίγον θέμα. Και επιτρέψτε μου ε, αρχικά δύο παρατηρήσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις και εκ μέρους της Επιτροπής και εκ μέρους του Frontex. Νομίζω οι δύο κύριοι απαντήσανε σε βάθος ερώτημα. Τον, η συζήτησή μας δεν αφορά τα μέτρα καταστολής όσον αφορά τους μετανάστες. Αυτό που ακούσαμε και από τους δύο κυρίους ήταν ε, μια υπαρίθμηση από μέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση των μεταναστών. Και αυτό το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο. Η συζήτηση γινόταν για την ε, βελτίωση, κατά τη γνώμη μου, για την ύπαρξη ανθρώπινων συνθήκων υποδοχής των μεταναστών. Και στο ζήτημα αυτό ούτε η Επιτροπή ούτε ο Frontex φυσικά, μπορούν να πούν οτιδήποτε γιατί εκπροσωπούν μια πολιτική που θεωρεί όπως αναφέρθηκε και ο συνάδελφος Μέγερ τους μετανάστες ως ε, εγκληματίες περίπου και φυσικά στη βάση αυτή έχουμε μόνον κατασταλτικά μέτρα. Ε, εμείς ήμασταν ούτως ή άλλως αντίθετοι με τη δράση του Frontex και από τα όσα είπε και ο κύριος ε, που την εκπροσωπεί σήμερα ε, δημιουργούνται πάρα πολύ σοβαρά ερωτηματικά και κάνω έκκληση σε εσά κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, να δούμε τη δράση του, του Frontex στην Επιτροπή μας και από τη σημερινή κατάθεση του κυρίου που ήταν μεταξύ μας. Ξέρουμε επίσης ότι η περιβόητη Task Force για τη Μεσόγειο αυτό που αποσκοπεί και είναι ρητή δήλωση είναι να αποτρέψει νέα κύματα μεταναστών να προσεγγίσουν τις ακτές της Μεσογείου. Αυτός είναι ο σκοπός της. Η Task Force Μεσόγειο θέλει την καταστολή των μεταναστών μπροστά στις ακτές της Αφρικής, όσο γίνεται πιο μακριά από εμά. Και ξέρετε κυρία Πρόεδρε, προέρχομαι από μια χώρα Προέρχομαι από μια χώρα όπου τα ζητήματα αυτά είναι πάρα πολύ έντονα, πολύ οξυμένα, οξύνονται κάθε μέρα και θα ήθελα με την ευκαιρία να αποκρούσω ένα επιχείρημα το οποίο έλεγε ότι ξέρετε όταν διευκολύνεται λέει τους μετανάστες γι' αυτό έρχονται και περισσότεροι στην, ε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράδειγμα της Ελλάδας δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, γνωρίζετε ότι η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής μεταναστών δεσμεύεται από τη συνθήκη του Δουβλίνου 2. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν από την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορούν να φύγουν από την Ελλάδα, δεν μπορούν, θέλουν να πάνε σε άλλες χώρες, δεν μπορούν να φύγουν η Ελλάδα έχει μηδαμινά ποσοστά παροχής ασύλου στους μετανάστες. Αυτά τα δύο πράγματα δεν έχουν εμποδίσει όμως χιλιάδες κυνηγημένους, εξατλειωμένους, πεινασμένους ανθρώπους και εξαιτία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις χώρες αυτές να, να αναζητούν ένα άλλο μέλλον ε, στην, ε, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κίνδυνο φυσικά τη ζωή τους ή αν θέλετε αντιμετωπίζοντας απαράδεκτες, απαράδεκτες από κάθε άποψη και το γνωρίζετε αυτό επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας που τους διώχνει πίσω κατά χιλιάδες αδιαφορώντας από πού προέρχονται. Απαράδεκτες συνθήκες κράτησης των μεταναστών στα διάφορα ε, νησιά του, ε, στην, στην, ε, στα, ελληνικά νησιά ή σε άλλες πόλεις. Έχουν μετατραπεί στρατόπεδα συγκέντρωσης που φιλοξενούν τους μετανάστες. Αυτά είναι τα ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα βάζει η, η, η, η συζήτηση που κάνουμε, αλλά σε αυτά δεν πήραμε καμία απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank Κυρία Χάουκεν, σας ευχαριστώ για την προσέλευσή σας. Όσο για την αναφορά, δεν ξέρω αν πρέπει να ευχαριστήσω για την απάντησή σας, γιατί το Frontex ακούγεται σαν ένα όργανο που δεν έχει κανένα μέσο αντίδρασης και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όσα προστάζει το διεθνές δίκαιο. Νομίζω ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα άμα συγκρίνουμε με άλλες γειτονικές δεν έχει ίδιο πρόβλημα. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχουν δραματικές καταστάσεις και δεν ανταποκρινόμαστε, δεν αντιμετωπίζουμε. Μιλάτε για μετανάστες που έρχονται από τη Συρία. Από ό,τι ξέρω εγώ, αυτοί ζητούν άσυλο και χρειάζονται προστασία. Και η πιο ευάλωτη ομάδα είναι οι Παλαιστίνοι από τη Συρία που αναγκάζονται να πάνε πρώτα στην Αίγυπτο όπου τους μεταχειρίζονται σαν εγκληματίες, τους φυλακίζουν και έχουμε και εδώ κάποια ευθύνη να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και όχι να τα αφήσουμε όλα όσα έχουν. Δύσκολο βέβαια για μας εδώ να κάνουμε τίποτε παραπάνω από το να αναγνωρίσουμε απλώς ότι υπάρχει τρομερό πρόβλημα που δεν το λύνουμε όπως θα έπρεπε. Πρέπει κάποτε να τα συζητήσουμε όλα αυτά πιο δημιουργικά. Καθώς και την έκθεση του διαμεσολαβητού γιατί εδώ ο καθένας αποφεύγει τις ευθύνες του, κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Και το Frontex γνωρίζει όπως και εμείς ότι ότι οι άνθρωποι αυτοί αν καταφέρουν να μην πνιγούν και παρά το ότι δεν μπορούν να φύγουν από την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία πάνε παρόλα αυτά θα συνεχίσουν να έρχονται. Βλέπετε τους αριθμούς. Και πρέπει να σεβαστούμε και το γεγονός ότι σε μερικές από τις χώρες προέλευσης τους γίνεται πραγματικά πόλεμος. Και είναι και αυτοί άνθρωποι σαν τους Ευρωπαίους. Και προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει ο κανόνας της Συμφωνίας του Δουβλίνου για να υπάρχει πιο μοιρασμένη ευθύνη Στη Δανία έχουμε πολύ λίγους μετανάστες γιατί μπλοκάρονται εκεί στις πρώτες χώρες όπου φτάνουν. How we Έχουμε βέβαια διαφορετικές αξίες ο καθένας και προοπτικές για τη ζωή του, αλλά αν θέλει κανείς να κατηγορήσει τη χώρα μου ότι δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της, σωστό θα ήταν Λόγω της νομοθεσίας όμως. Γιατί ξέρουμε ότι δίπλα μας συμβαίνουν, σημειώνονται τρομακτικοί πόλεμοι. Αλλά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αυτοί είναι αιτητές ασύλου και όχι απλώς παράνομοι μετανάστες. Ευχαριστούμε κύριε Χάουκεν, ο κύριος Αλαβράκος. Ευχαριστώ κύριε. Danke Και τους άλλους αναφέροντες από το σημείο 6 μέχρι το 13, οι οποίοι θέτουν τα κεφάλαια της ουσιαστικής αντιμετώπισης της μεταναστευτικής πολιτικής. Ε, άκουσα με πολύ προσοχή την Κομισιόν. Μας αναφέρθηκε ε, σε ένα νομικό καθεστώς του Δουβλίνου 2 δεν μπορούσε τίποτα άλλο να κάνει. Άκουσα τη Frontex και με ε, επενετή ε, κατά κάποιο τρόπο ε, συμπεριφορά ενώπιόν μας είπε ότι ο ρόλος μας είναι συντονιστικός έχουμε μικρές δυνάμεις και απλούστατα αποκτάμε μια εμπειρία. Το ρόλο αυτό της Frontex εγώ τον χαιρετίζω. Τον χαιρετίζω διότι για πρώτη φορά δια της ιδρύσεως της ΦΟΔΕΣ και της Tax Force αναγνωρίσαμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά σύνορα και επομένως το μεταναστευτικό είναι ευρωπαϊκό θέμα. Διότι ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση δεν έχουμε. Το θέμα του πολιτικού ασύλου. Το θέμα του πολιτικού ασύλου είναι άλλο και είναι πολύ πιο μικρό από ό,τι είναι το μεταναστευτικό. Να πω χαρακτηριστικά ότι στην Ελλάδα έχουμε 16.000 αιτήσει ε, παροχές πολιτικού ασύλου, εκ των οποίων έχουν ικανοποιηθεί περίπου οι πέντε. Έχουμε όμως 1,5 με 2 εκατομμύρια μετανάστες. Αντιλαμβάνεστε ότι το μέγεθος σε σχέση με τον αριθμό των μεταναστών και τον αριθμό των ετούντων άσυλο είναι πάρα πολύ μικρό. Πέρυσι κάηκε ε, ένα εργοστάσιο στο Μπαγκλαντές. Στο Μπαγκλαντές κάηκαν 137 παιδιά ηλικίας από 8 έως 14 ετών που δούλευαν στο εργοστάσιο αυτό για 37 δολάρια το μήνα. Είπα τότε ότι μία από τις αιτίε που φεύγει ο κόσμος και έρχεται προς την Ευρώπη είναι και το οικονομικό. Είπα να πάρουμε μέτρα και να καθορίσουμε ένα παγκόσμιο κατώτατο μισθό. Να πούμε 150 δολάρια. Αν τους δώνουμε 150 δολάρια εκεί, εν πάση περιπτώσει, σαν εργατική νομοθεσία θα μπορέσουμε να κρατήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι. Βεβαίως αυτό είναι αντίθετο σε πολλά συμφέροντα και ουδής το ακολούθησε διότι ε, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι και η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με άλλα κράτη οφείλεται στο γεγονός ότι γίνεται εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και οι παρενέργειες αυτή της εκμετάλλευσης είναι ότι έρχονται σαν μετανάστες στην Ευρώπη για μια καλύτερη τύχη. Ε, Εκείνο το οποίο ε, θα πρέπει να δούμε είναι ότι καθίσαμε στο Δουβλίνο 2, καθορίσαμε τις ε, χώρες χωματερές, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, είπαμε εκεί τους πετάμε όλους και έληξε η ιστορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα με το πρόβλημα της Λαμπεντούσας ε, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι ότι για χίλιους μετανάστες τα κράτη του Βορρά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν το χατήρι για χίλιους μετανάστες να δεχθούν το Λουξεμβούργο παραδείγματος χάρη 10 η, Δανία 45 ε, η Γερμανία κάπου 150 και λύσαμε το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. ή πρέπει να αναμορφώσουμε την πολιτική εάν είναι για χίλιους ανθρώπους να ευγνωμονούμε τα βόρεια κράτη επειδή τα παίρνουν και να μας αφήνουν τα εκατομμύρια στην Ελλάδα και στην Ιταλία τότε αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για άλλου είδους αλληλεγγύη. Μια αλληλεγγύη αλλά κάρτα. Ένας από τους λόγους για τους οποίους πρέπει να αντιληφθούμε ότι η μετανάστευση πρέπει να πάρει μια μορφή ευρύτερης σχεδιάσεως είναι και το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Άρα τουλάχιστον 50 εκατομμύρια μετανάστες μέχρι το 30 πρέπει να τους κάνουμε Ευρωπαίους πολίτες. Και πώς θα τους κάνουμε Ευρωπαίους πολίτες. Με τον τρόπο αυτό, έχοντας τους παράνομους σε κάθε χώρα, οθώντας τους με αυτόν τον τρόπο ε, στην παρανομία και την παντός είδους εκτέλεση αξιοπίνων πράξεων εάν δεν μπορέσουμε να τους απορροφήσουμε μέσα στον ιστό της Ευρώπης, αντιλαμβάνεστε ποια θα είναι η Ευρώπη του 2030. Θα έχουμε ένα γυρασμένο ευρωπαϊκό πληθυσμό και τους νέους αυτούς ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στην παρανομία. Ή οι περισσότεροι από αυτούς θα είναι στην παρανομία. Προέχει η άποψη του αναφέροντος και η πρόταση του αναφέροντος ότι πρέπει να γίνει ένα συντονιστικό συμβούλιο είναι το πρώτο το οποίο αν θέλουμε να μιλάμε ουσιαστικά πρέπει να προωθήσουμε. Ένα ουσιαστικό ε, συμβούλιο το οποίο τι θα κάνει, θα κάνει τις ποσοστώσεις. Κάθε χώρα πρέπει να δεχθεί έναν αριθμό ανθρώπων οι οποίοι μεταναστεύουν. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Δεν μπορούμε αλλιώς τη μετανάστευση με τις απαγορεύσεις να την κρατήσουμε και από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στην Ελλάδα να έχει μεταναστευτικά εμβάσματα 9 δισεκατομμύρια το μήνα, το, χρόνο και 30 δισεκατομμύρια τα τελευταία πέντε χρόνια και να λέμε «Α, οι Έλληνες είστε και απαταιώνες και φάγατε τα λεφτά». Μα δεν είναι έτσι. Αποδομούνται οι δομές. Αποδομούνται οι δομές της Ιταλίας. Μπορεί είναι η Ελλάδα με 10 εκατομμύρια πληθυσμό να αντέξει 20% παραπάνω πληθυσμό που θέλει σχολείο, θέλει νοσοκομείο, θέλει όλες αυτές τις δυνατότητες που χρειάζεται ένας άνθρωπος, εκτός αν θέλουμε να τους κάνουμε υποζύγια. Δεν είναι στην παιδεία ούτε στην κουλτούρα των Ελλήνων να τους κάνουν υποζύγια. Όμως υπάρχουν εξαρτήσεις και οι εξαρτήσεις βλέπω ότι ε, γίνονται από πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα και φοβάμαι και αλλού Ορισμένες από αυτές εμφανίζονται και πολύ αριστερές μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες εκμεταλλεύονται τον πόνο αυτών των ανθρώπων και την αδυναμία αυτών των ανθρώπων να εμφανιστούν σαν άνθρωποι. Κρύβονται. Κρύβονται σαν σκυλιά στους δρόμους γιατί δεν έχουν τα ένταφα. Ε, λοιπόν, αυτή είναι η προοπτική που δίνουμε στη μετανάστευση. Και θα το συζητήσουμε εδώ και θα λήξει το θέμα. Θα πάμε στα γραφεία μα και θα πούμε «Α, είπαμε ο καθένα πέντε κουβέντε ωραίε Και από εκεί και ύστερα έλειξε το θέμα το μεταναστευτικό. Διότι αυτό βλέπω και γίνεται. Κουβεντούλε κάνουμε. Κουβεντούλε και δι υποκριτικέ κουβεντούλες. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, γιατί για το θέμα αυτό μπορεί κανεί να μιλήσει επί πέντε ώρε Τουλάχιστον πρέπει να αποφασίσουμε ότι δεν υπάρχει Δουβλίνο 2 και πρέπει να χαράξουμε μεταναστευτική πολιτική. Το θέλουμε, θα το δείξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Mr. Ja, vielen Dank, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich finde es erstmal außerordentlich. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι συζητάμε το πρόβλημα και από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και εύκολη η λύση. Εγώ λοιπόν θέλω να παρακαλέσω να είμαστε ειλικρινείς, να τα πούμε ξεκάθαρα μεταξύ μας. Ε, θα πω κι εγώ κάποια πράγματα που με απασχολούν. Βεβαίω και μπορεί κανείς να πει ότι η μεταναστευτική πολιτική ή αν θέλετε οι χειρισμοί των ετούντων άσυλο είναι καθαρά ευρωπαϊκό καθήκον. Και εκεί η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη. Σωστά το είπατε. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να σας πω το εξή. Πρέπει κανείς να θέσει το εξή ερώτημα. Πώς θα τα οργανώσουμε όλα αυτά, γιατί χωρίς κανόνες δεν γίνεται και κάποια στιγμή, ακόμα και με αλληλεγγύη, τίθεται το ερώτημα σε τελική ανάλυση Πόσους ετούντες άσυλο μπορεί να δεχτεί αυτή η Ευρώπη. Ένα εκατομμύριο, δύο, εκατό εκατομμύρια. Έρχονται μετά και άλλοι και λένε χρειαζόμαστε νόμιμη μετανάστευση. Τι ακριβώς εννοείται με νόμιμη μετανάστευση. Δηλαδή θα κάνουμε επιλογή και θα παίρνουμε τους καλύτερους. Αυτοί που είναι καλά εκπαιδευμένοι, αυτοί να έρχονται. Οι άλλοι χάσανε να μείνουν απ' έξω. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση και να την κάνουμε ευθύ εξ αρχή. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος θα μπορούσε να είναι αγγελικά πλασμένος, αλλά δεν είναι. Στη Γερμανία, ας πούμε, 100 ε, ευρώ το μήνα δίνουμε εμεί σε κάθε από αυτού του μετανάστε και αυτοί τα 100 ευρώ δεν έχουν τίποτε στη ζωή του. Το καταλαβαίνω λοιπόν ότι θέλουν να έρθουν σε εμά. Και να πω και κάτι άλλο για τη Frontex. Δεν πρέπει να ζητάμε από τη Frontex πράγματα για τα οποία δεν είναι αρμόδια Frontex. Διότι η Frontex, ε, ξέρετε, ε, φτάνει σε καθυστερημένη φάση μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν έχει αποτύχει η εξωτερική πολιτική και η αναπτυξιακή πολιτική και έρχονται οι άνθρωποι αυτοί πια σε έδαφος της Ευρώπης, τότε είναι πολύ αργά. Κάτι δεν πήγε καλά. Γιατί, διότι οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να έρθουν σε εμά όπως είπατε, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. Το μόνο που μπορεί να κάνει Frontex είναι να διαχειριστεί την καταστροφή. Αυτό μπορεί να κάνει. Και το κουβεντιάζουμε και αυτό αν θέλετε. Επίσης, θα επιθυμούσα να πάρουμε και την ειδική έκδοση της διαμεσολαβήτριας. Βεβαίω και το πρόβλημα είναι πολυπίπεδο και εγώ το καλό θέλω, αλλά ξέρετε δεν είναι εύκολο να απαντηθεί το ερώτημα, δεν είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια εκτεταμένη συζήτηση και ειδικά στη Frontex που δέχεται τόσο έντονη κριτική Θέλω να προσθέσω, δεν μπορούμε να επιλέγουμε ένα στοιχείο και να επιτιθέμεθα με βάση αυτό. Τα προβλήματα είναι πολλά, είναι πολύ επίπεδα, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Και να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως, εκ των υστέρων πολλά μπορεί κανείς να εξηγήσει, αλλά ε, θα θυμάστε όλοι μας ήμασταν κατενθουσιασμένοι με τον εκδημοκρατισμό της Βορειοαφρική και λέγαμε επιτέλους δημοκρατία. Αυτό ήταν η μία πλευρά του νομίσματος και η άλλη πλευρά όμως είναι ότι οι πρόσφυγες, ο αριθμός τους αντί να μειωθεί αυξήθηκε. Κάτι λοιπόν δεν πάει καλά. Άρα πρέπει να συζητήσουμε και γι' αυτό. Και τελειώνοντας να σας πω ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για αυτό το δύσκολο πρόβλημα. Ο κύριος Μποστινάρου τελευταίος. Κύριε Πρόεδρε, Χωρίς να προσθέτω τίποτε ουσιώδες παραπάνω, θα ήθελα να θυμίσω ότι πρώτον είναι βασικό να έχουμε την έκθεση του διαμεσολαβητή για το Frontex. Δεύτερον, επαναλαμβάνω την έκκλησή μας να γίνει μία γνωμοδότηση για αυτό το θέμα, καιρός είναι επιτέλους και τέλος μην ξεχνάτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο να αρχίσει την προετοιμασία μιας νέας ενωσιακής πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση. Και τα κράτη-μέλη ακόμη αντιτίθενται και το συζητάνε. Γι' αυτόν τον λόγο τελικά στο τέλος της Φιλανδικής Προεδρίας μας είχαν υποσχεθεί ότι θα υπάρξει μια πραγματική επιτέλους ενωσιακή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου, αλλά πόρο απέχει ακόμα με τη Λαμπεντούζα. Φάνηκε μόνο το μέγεθος της τραγωδίας. Υπάρχουν και πολλές αναφορές για αυτά τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου και το πρόβλημα γίνεται όλο και σημαντικότερο και δραματικότερο και καθήκον μας είναι ως Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να γνωμοδοτήσουμε γιατί εγκαίρως, γιατί μετά τις εκλογές θα χρειαστεί ακόμα πιο πολύ να αλλάξει η ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε συνεχώς τραγωδίες σαν τις Λαμπεδούσεις σαν να είναι κανονικές. Ο κύριος Φρατέλο για μία μονόλεπτη απάντηση. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ε, πλούτησαν τη συζήτηση με τις παρεμβάσεις τους, τους βουλευτές κυρίως, αλλά και τη Frontex. Ε, βλέπω ότι παρακολουθείτε με προσοχή αυτή την αναφορά Αναφερθήκατε στις δραστηριότητες τις οποίες έχουν ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες, οι οποίες όμως έχουν ε, στόχο θα έλεγα βραχυπρόθεσμο. Το θέμα είναι ε, εκ των προτέρων να λύνουμε τα θέματα, να τα προλαμβάνουμε. Ε, εν πάση περιπτώσει θα πρέπει η Ευρώπη να κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το θέμα είναι τι δράσεις μπορούμε να αναλάβουμε μακροπρόθεσμα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το καθεστώς της μετανάστευσης στη Μεσόγειο, όχι μόνο για να ασκήσουμε κριτική, αλλά σε οργανωτικό επίπεδο. Εκ των κάτω θα πρέπει να δούμε τι λύσεις προτείνονται τοπικά και πώς μπορούμε όλες αυτές τις λύσεις να τις προσθέσουμε και να συνεργαστούμε με τους πρωτογονιστές του συγκεκριμένου φαινομένου και έτσι θα προσφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιμετώπιση αυτού του δύσκολου προβλήματος. Νομίζω ότι ε, είναι απαραίτητο βέβαια και κάποιες δράσεις βραχυπρόθεσμες ε, να αναλυθούν προσπάθειες όπως ε, ο περιορισμός του αριθμού των, θα έλεγα, των μεταναστών να μην ξεκινούν εύκολα, να μειωθεί φυσικά ο αριθμός των θυμάτων δεν μπορούμε φυσικά να σταματήσουμε τα μεταναστευτικά ρεύματα. Αυτό η ιστορία δείχνει ότι δεν μπορεί να γίνει, αλλά να τα ελέγξουμε με κάποιο τρόπο. Σας ευχαριστώ λοιπόν γιατί μας παρουσιάσατε ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο εξ ονόματος όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στράφηκαν στην Επιτροπή μας γύρω από το συγκεκριμένο θέμα προέρχονται από διάφορες χώρες, όπως είπα στην ανακοίνωση των αναφορών, έχουν κατατεθεί από Αυστριακούς, Έλληνες, Γερμανούς, δείχνουν ότι το θέμα το οποίο μας απασχολεί σήμερα δεν είναι κάτι το οποίο αρχίζει και τελειώνει στη Λαπεντούσα. Όπως και εσείς ο ίδιος είπατε, το θέμα δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ε, μόνο όταν γεμίσει πτώματα η μεσογειακή λεκάνη, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί με οργανωμένο τρόπο, με συντονισμό και στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής λογικής, μιας κοινοτικής λογικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του εκπροσώπου της και σήμερα ε, μας ε, έδωσε ακριβώς τη σημασία που έχουν οι εθνικές παρεμβάσεις περισσότερο παρά οι ευρωπαϊκές. Είναι αλήθεια ότι έχουν ξεκινήσει αρκετές πρωτοβουλίες ε, μετά από πιέσεις κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέσω των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έχουμε πιέσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν και έχει θέσει αν θέλετε σε δράση και αναπτύσσει αυτή τη στιγμή κάποια μέσα. Μέσα τα οποία αντιπροσωπεύουν κάποια μεμονωμένα μικρά βήματα τα οποία σίγουρα δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσουν την συντονισμένη προληπτική δράση πριν εξελιχθούν τα φαινόμενα και πριν τρέχουμε συστηματικά πίσω από τα γεγονότα. Είναι λοιπόν σαφές ότι η συγκεκριμένη αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή διότι το πρόβλημα δυστυχώς παραμένει χένον. Είναι ε, κάτι το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει ε, σε ιστερότερη φάση να αναζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερα στα πλαίσια της προοπτικής ε, ε, εισαγωγής νέων νομοθετικών μέτρων ευρωπαϊκού επίπεδου που ορίζουν θέματα όπως η χορήγηση ασύλου, τα δικαιώματα των προσφύγων, η απόδοση μιας προοπτικής σε κάποιους ανθρώπους όπου αυτό είναι απαραίτητο, γιατί αν δεν φτάσουμε σε μια τέτοια ευρωπαϊκού επίπεδου λύση θα το αντιμετωπίζουμε πάντα με μια διασπορά πόρων, όχι μόνο οικονομική αλλά κυρίως ανθρώπινη. Ε, μιλάμε για πολίτες οι οποίοι θέλουν να ζήσουν, θέλουν τα δικαιώματά τους να γίνουν σεβαστά και προσβλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να φτάσουν σε αυτή. Λοιπόν κλείνοντας να πω ότι παραμένει ανοιχτή η αναφορά. Θα ζητήσω από τους συντονιστές να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα έτσι ώστε να καθοριστεί και από πλευράς δικής μας μια πιο συγκεκριμένη στρατηγική έτσι ώστε να μην συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα να λέμε λόγια και να μην κάνουμε πράξεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας όλους εδώ. Κλείνω το συγκεκριμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Περνώ τώρα στο επόμενο θέμα. Πρόκειται για την αναφορά την οποία έχει καταθέσει ο Τζουζέπε Λαμπαρέλη, ο οποίος έχει αποστείλει ένα σημείωμα με διευκρινήσεις το οποίο διανεμήθηκε μόλις τα μέλη της Επιτροπής για να αντικαταστήσει την παρουσία του εδώ. Έχει σαν στόχο λοιπόν την μεταρρύθμιση των τοπικών αρχών που έχει ξεκινήσει στην Ιταλία. Σύμφωνα με τον αναφέροντα είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα στις εδαφικές ισορροπίες οι δράσεις τις οποίες θέλει να αναλάβει η κυβέρνηση της Ιταλίας είναι αντίθετη με την αρχή την οποία προβλέπει το άρθρο 1 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, ε, οδηγεί στην δημιουργία μιας ένωσης στενής ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες με πιο ε, διαφανή τρόπο ε, για τον Ευρωπαίο πολίτη. Η διατύπωση των ε, αναφερόντων καταγγέλουν τη συμπεριφορά της ε, Ιταλικής κυβέρνησης γιατί παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα που βρίσκονται στα θεμέλια της ίδιας της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα άρθρα 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21 και 41 που αφορούν την απονομή δικαιοσύνης, την χρηστή διαχείριση ε, και άλλα δικαιώματα και υπάρχουν ε, λοιπόν και άλλα δικαιώματα που παραβιάζονται. Συμμετέχουν επίσης ε, εκπρόσωποι διαφόρων τοπικών Ιταλικών αρχών που θέλουν και αυτοί να τονίσουν ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης τον μήνα Μάρτιο αμφισβήτησε ε, τις Ιταλικές αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο αγνόησαν τις απόψεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε σχέση με το άρθρο 315 του κανονισμού λειτουργίας των περιφερειακών και τοπικών αρχών σε σχέση με τις προμήθειες των Δήμων και Κοινοτήτων όπως επίσης και το θέμα της εκλογής των περιφερειακών και επαρχιακών αρχών στη συγκεκριμένη χώρα. Σε 19 από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν τρία επίπεδα διακυβέρνησης. Μόνο κάποιες μικρές χώρες όπως η Κύπρος, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο δεν διαθέτουν επαρχιακές αρχές. Τα δικαιώματα λοιπόν των αρχών των Ιταλικών επαρχιών σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών παραβιάζεται από τις προτάσεις της Ιταλικής κυβέρνησης. Οι γερμανικές επαρχίες για αυτές τις υπηρεσίες διαχειρίστηκαν 55 δις τον προηγούμενο χρόνο, 73 δις οι γαλλικές επαρχιακές αρχές και οι ιταλικές πόσα κάτω των 10. Συνεπώς λοιπόν οι ιταλικές επαρχίες δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο το 1,26% του κρατικού προϋπολογισμού της χώρας. Λοιπόν, η πρόταση της Ιταλικής κυβέρνησης δεν μπορεί να είναι η απάντηση ε, για μια σωστή εξοικονόμηση πόρων στους εθνικούς προϋπολογισμούς γιατί κάτι τέτοιο θα παραβιάσει τα αναλύωτα δικαιώματα των χωρών και των πολιτών. Συνεπώς λοιπόν ε, θα πρέπει να δούμε σύμφωνα με την αναφορά όχι μόνο τις συγκεκριμένες αποφάσεις της Ιταλικής κυβέρνησης για την αναδιάταξη των Ιταλικών επαρχιών αλλά και τις αιτίες οι οποίες οδήγησαν στην συγκεκριμένη αυτή αλλαγή. Όπως είπα ο αναφέρον δεν είναι παρόν και θα δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι δικαίωμα του κάθε κράτους μέλους ε, να ανακοινώνει μόνο του τις οργανωτικές δομές, ότι δεν υπάρχει εδώ ε, ευρωπαϊκή αρμοδιότητα σύμφωνα με τη συνθήκη. Και κανένα άλλο σχόλιο. Πάρα πολύ ωραία, λέει η Πρόεδρος. Μήπως θέλει κάποιος ε, να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. δεν μπορώ εγώ να συμφωνήσω με την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν η ίδια μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι δεν μπορεί να μπει σε θέματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτέτων ε, της ε, κυβέρνησης και της κυβερνητικής διοίκησης κάθε χώρας ακόμα και σε σχέση με θέματα που αφορούν την αυτονομία των επαρχιών και των, επαρχιακών, περιφερειακών και τοπικών αρχών. Βέβαια η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεκδικεί παρέμβαση στον τομέα σαν παράδειγμα του εργατικού δικαίου, των ρυθμίσεων για την προστασία των εργαζομένων κτλ. που δεν είναι κανονικά θέματα που εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα θέματα βέβαια της οργάνωσης των περιφερειακών και τοπικών αρχών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει τον πόντιο πιλάτο. Και όταν λένε τέτοια πράγματα οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αντιμετωπίζονται πάρα πολύ αρνητικά σε περιοχές όπως ε, η ε, Καταλωνία. Όταν άπτεται λοιπόν των θεμάτων ε, που αφορούν τις περιφέρειες και τους λαούς ε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση της δικής μου χώρας ε, πρέπει να γνωρίζει ότι η κοινωνία υποστηρίζει κάποιες μεταρρυθμίσεις και δεν μπορεί να λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για την Ιταλία. Νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη αναφορά οι Ιταλοί πολίτες θεωρούν ότι θα πρέπει οι περιφερειακές αρχές να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις γιατί είναι κοντά ε, στους ε, πολίτες και υπάρχουν πολύ σημαντικές μορφές ε, οργάνωσης περιφερειακής και γι' αυτό είναι σε θέση να εντοπίσουν τα προβλήματα τα οποία έχουν μπροστά τους οι Ευρωπαίοι πολίτες με τη σωστή εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας ανάμεσα σε άλλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο κ. Μποστινάρου. Έχοντας ακούσει τις δηλώσεις τις οποίες έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας μόνο το εξής Κάθε κράτος μέλος είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφασίζει για την δική του εθνική μορφή διοικητικής οργάνωσης. Πρώτον ήταν αυτό. Δεύτερον, κάθε αλλαγή στα πλαίσια των συνταγματικών ορίων και αρμοδιοτήτων είναι θέματα που αφορούν την αρχή της επικουρικότητας ελέγχεται μεν ο προϋπολογισμός εκ των προτέρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να εκπληρεί συγκεκριμένα κριτήρια ε, στον τομέα της μακροαιρεσιμότητας κτλ. Αλλά ποτέ, ίσως να κάνω λάθος, διορθώστε με, αλλά ποτέ δεν μπαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, κατανομή λεπτομερώς των διαθεσίμων πιστώσεων προς τις επαρχίες, τους δήμους, τις κοινότητες και τις επαρχίες γενικότερα. Το μόνο θέμα λοιπόν το οποίο τίθεται όπως και εσείς ε, μας ζητήσατε είναι σαν μέλος της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων. Ο μόνος τομέας στον οποίο έχει κάτι να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο ρόλος ε, των διαχειριστικών λεγόμενων αρχών. Εφόσον υπάρχει λοιπόν ε, ε, περιφερειακό επίπεδο λήψης αποφάσεων, τότε θα πρέπει με διαχειριστικές ικανότητες των κοινοτικών ταμείων κτλ. θα πρέπει εκεί να περνάει από διαδικασία ελέγχου από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέραν τούτου ουδέν. Και το θέμα αυτό αφορά την Ιταλία και δεν αφορά την Καταλωνία συνάδελφε. Και καλό είναι να μην ανακατεύουμε πράγματα τα οποία είναι ανώμια εν πάση περιπτώσει και γι' αυτό και εγώ θα ζητήσω η συγκεκριμένη αναφορά να κλείσει. Η κυρία Ούκεν. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω δανέζικα. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής. Θυμάμαι, ήμασταν στη Ρώμη και εκεί συζητεί το, το θέμα τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα και αυτό που πραγματικά ήταν εντυπωσιακό ήταν ότι υπάρχουν ε, ε, πάρα πολλά διοικητικά επίπεδα, δήμαρχοι και άλλοι πολλοί οι οποίοι ε, μετακυλίουν τις ευθύνες ο ένας τον άλλον. Και τελικά κανείς δεν έφερε την ευθύνη για τα απόβλητα. Στην προεκλογική λοιπόν εκστρατεία ο Υπουργός είπε ότι πρέπει αν θέλει να λάβει μια απόφαση να απευθυνθεί σε 561 δημάρχους. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν γίνεται τίποτα ούτε και στους μικρούς δήμους και μετά υπάρχουν και οι μεγάλοι δήμοι. Νομίζω λοιπόν ότι το σύστημα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Αυτό όμως δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο, ε, με κάθε σεβασμό κυρία Πρόεδρε, απευθύνομαι στον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν και λέω ότι κάτι πρέπει να κάνει. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Μου κάνει εντύπωση ε, που έγινε δεκτή αυτή η αίτηση, ενώ έχουμε απορρίψει πάρα πολλές άλλες που θα έπρεπε να τις δεχτούμε και τώρα αυτό που είναι γενικό και περί Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέτοια, αυτό το δεχτήκαμε. Ε, δεν καταλαβαίνω καλά το συνάδελφο. Ευτυχώς ε, βέβαια είμαι σε διαφορετικές <laughs> πολιτικές ομάδες, αλλά διαφωνούμε. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτό δεν πρέπει να το δεχτούμε ως ε, αναφορά. Δεν μπορώ να φανταστώ ποια λύση μπορούμε να βρούμε σε αυτό το πρόβλημα. Κατανοώ πολύ καλά τη στάση της Επιτροπής και με μεγάλη μου χαρά συμμετέχω στη συζήτηση για το πώς μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος, αλλά νομίζω δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα για αυτό το θέμα. Να το κλείσουμε το θέμα και τέλος. Παρακαλώ, ο κύριος Γιάρ. Κοιτάξτε, η δική μου η πολιτική ομάδα θεωρεί ότι θα πρέπει κανείς να δέχεται και την αντίθετη άποψη. Εγώ λέω να την αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να τη συζητήσουμε. Να δούμε τι θα κάνουμε. Κοιτάξτε κυρία ε, Χοκ, ε, προηγουμένως συμφωνήσαμε μια φορά φτάνει, δεν γίνεται, ε, φτάνει και ήταν και πολύ. Δυστυχώς οι παρατηρήσεις λέγονται, γίνονται εκτός μικροφώνου. Πρόεδρος, αυτά που ακούμε σήμερα είναι πράγματι πρωτοφανή. Για δεύτερη φορά φαίνεται ότι συμφωνεί η κυρία Χόκεν με τον συνάδελφο κύριο Γιάρ και εδώ ε, θέλω να προσθέσω, εσείς ζητήσατε να κλείσει, όχι, από τη μετάφραση κάποιο πρόβλημα προέκυψε. από ό,τι κατάλαβα ζητήσατε να κλείσει. Τέλος πάντων, ε, προέκυψε κάποια παρεξήγηση. Ε, από ό,τι φαίνεται όμως δεν συμφωνείς τελικά. κακός είπα εγώ ότι συμφωνήσατε. Δεν επικράτησε αυτό το κλίμα των Χριστουγέννων. Νομίζω ότι θα πρέπει να τοποθετηθούμε με ψηφοφορία. Ψηφιστικός. Ο κύριος Γιάρ εκπροσωπεί το ΕΛΚ, ο κύριος Μποστινάρου του Σοσιαλιστές. Αλλά ας πούμε οι πράσινοι είναι διχασμένοι. Πρέπει λοιπόν να καταφύγουμε στην ε, ψηφοφορία. Κοιτάξτε, αν κάποιος θέλει να παραμείνει ανοιχτή, ας την κρατήσουμε ανοιχτή. Αυτή την αρχή εφαρμόζω εγώ εδώ. Αν ο Πέτρος Γιάρα θέλει να δοθεί ιδέουσα απάντηση και τα λοιπά, θα με ενδιαφέρει και εμένα, γιατί όχι. Ευχαριστούμε κυρία Χάουκεν. Δέχεστε την πρόταση της κυρίας Χάουκεν λοιπόν. Α, μάλιστα. Θα κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή και θα ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Τώρα το 16. Το 16. Η αναφορά της Αντάστρα μια ένωση Ρουμάνων επιστημών σχετικά με καζόμενη παραβίαση τη κοινωτική νομοθεσία σχέση με το έργο κατασκευή χρυσοργείου στη Ρώσια Μοντάνα στη Ρουμανία. Μαζί με την αναφορά του Σόριν Γιούρκα για το ίδιο θέμα και την αναφορά ενός Ρουμάνου πολίτη για το ίδιο θέμα. Ένας από τους αναφέροντες είναι εδώ. ο κύριος Οκτάβιος Γουικουλέσκου εκ μέρους της Αντάστρα. Μπορεί να μιλήσει επί πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω την αναφορά μας και γιατί κρατήσατε το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είναι πολύ επίκαιρο γιατί δεν υπήρξε καμία πρόοδος για κανένα από τα θέματα που συζητήθηκαν. Αντίθετα υπάρχουν νέα στοιχεία που ενδυναμώνουν τις αμφιβολίες μας για αυτό το θέμα. Ίσως να γνωρίζετε ότι το θέμα της Ρώσια Μοντάνα ε, άρχισε να ενδιαφέρει ολόκληρη την κοινωνία και εξόργησε ορισμένους δημιούργησε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στη χώρα εδώ και 23 χρόνια. Επομένως, ο διχασμός και οι συζήτηση αυτές δείχνουν το ενδιαφέρον των πολιτών. Θα θέλαμε λοιπόν να δηλώσουμε εκ νέου ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πρόγραμμα αυτό, να γίνουν ανεξάρτητες αξιολογήσεις και Απαιτείται βέβαια και η εφαρμογή της αρχής της φρόνησης, όπως λέει το άρθρο 191 της συνθήκης. Αυτό το θέμα μοιάζει αρκετά με αυτό που ακούσαμε μόλις παρα προηγουμένως. Να σας κάνω, αναφέρω τα κυριότερα προβλήματα. Το πρόγραμμα είναι πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων από οποιοδήποτε ανάλογο στην Ευρώπη είναι δύσκολο να καταλάβει καλή στην κλίμακά του. Βάσει των αριθμών που δίνει η εταιρεία η ίδια, το κέρδος από, για το Ορμανικό κράτος θα αντιπροσωπεύει περίπου το βάρος ενός δαχτυλιδιού, χρυσού δαχτυλιδιού αλλά θα δημιουργήσει 10 τόνους αποβλήτων 8 κυβικά μέτρα για κάθε μονάδα. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπου υπάρχουν και πολλά προστατευόμενα είδη πουλιών και ζώων. Τα ύδατα που θα δημιουργηθούν για τον καθαρισμό θα κρατιούνται από ένα φράγμα 1350 μέτρων μήκους. Αυτό σας δείχνει πόσα πολλά απόβλητα θα δημιουργηθούν. Από περιβαλλοντολογικής απόψεως η εταιρεία μας έδωσε ένα χάρτη όπου δεν εμφαίνεται κανένα γεωλογικό σφάλμα ή ρήγμα. Αλλά ο χάρτης αυτός διαφέρει από έναν χάρτη του 70 τον οποίο μπορέσαμε να βρούμε αρκετά εύκολα από το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ρουμανίας, όπου βλέπουμε δύο κύρια ρήγματα, όπου θα κρατούν τα ύδατα. Σε κλίμακα 1 προς 50.000 είναι φανερά αυτά τα ρήγματα. Επομένως πρέπει να γίνει μια πιο ενδελεχής έρευνα γεωλογική. Δύο κορυφαίοι επιστήμονες στο Γεωλογικό Ινστιτούτο ε, ήρθαν στη Βρετανική Βουλή και επιστοποίησαν τη γνησιότητα αυτών των χαρτών. Έχω αντίγραφά τους εδώ και των δύο, και του Γεωλογικού Ινστιτούτου και της εταιρείας. και μπορούμε πολύ εύκολα να πάρουμε αντίγραφα από το Γεωλογικό Ινστιτούτο. Αυτό φυσικά αμφισβητεί την αξιολόγηση του κινδύνου που έγινε από την εταιρεία. η οποία βέβαια έχει και το άχθος της αποδείξεως για τις κατηγορίες μας. Μας λέει απλώς ότι είναι ανυπόστατα αυτά που λέμε και ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν καμία αλλαγή. Οι χρηματικές εγγυήσεις που δίνει η εταιρεία δεν έχουν καμία σχέση με το πραγματικό πρόβλημα. Έχει προβλεφθεί αποζημίωση 10 φορές μικρότερη από ό,τι σε ανάλογες περιπτώσεις, αν υπάρξει ατύχημα, πληρώθηκε λένε ότι είναι πάρα πολύ ασφαλείς οι εγκαταστάσεις και γι' αυτό προβλέπεται τόσο χαμηλή αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος. Φέτος όμως μία μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία αρνήθηκε να ασφαλίσει το πρόγραμμα. Και δεν υπάρχει καμία λεπτομέρεια ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης πιθανών ατυχημάτων και το κόστος. Η αρχή της φρόνησης λοιπόν και με βάση το άρθρο 2 απαιτεί να εφαρμοστεί η οδηγία του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορά αυτά τα τέτοιου είδους εγκαταστάσεις πριν εγκριθεί το σχέδιο. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δείχνει ότι στο μέλλον δεν αρκούν τα προβλεπόμενα μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος, αλλά χρειάζονται πολύ σοβαρότερα. Εδώ θα καταστραφεί σχεδόν ολόκληρος ο αρχαιολογικός χώρος που υπάρχει εκεί και όταν θα σκαφτεί το βουνό που όπως προβλέπει η εταιρεία. Ενώ έχει ζητηθεί επανειλημμένως η συντήρηση του χώρου αυτού Πρόσφατα ακαδημαϊκοί από την Οξφόρδη και το Λέστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο δημοσιεύτηκαν μελέτες που είχε παραγγείλει η κυβέρνηση από το 12 όπου οι ακαδημαϊκοί λένε ότι ο αρχαιολογικός χώρος είναι πολύ μεγάλης παγκόσμιας αξίας και μπορεί να εγκριθεί και ως παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO και ζητούν και αυτή τη διατήρησή του. Η Ευρώπη λέει ότι προστατεύει την πολιτιστική κληρονομιά ενώ παράλληλα καταστρέφονται τέτοιοι χώροι. Ευχαριστώ. Η καταστροφή του χώρου αυτού λοιπόν θα είναι μεγέθους που δεν έχει φανεί στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Προβλέπεται να σκαφτούν σύραγγες τεράστιες που μόνο στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχαμε δει να σκάβονται. Δυστυχώς βέβαια δεν έχουμε τα αρχεία των προγόνων μας για να ξέρουμε πώς αντιμετώπισαν εκείνοι, εκείνα τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πάρει και άλλες αναφορές γύρω από το θέμα, αλλά και για διάφορες χώρες και για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Θα δώσω το λόγο τώρα στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε για το θέμα της Ρώσια Μοντάνα. Έχουμε λάβει λοιπόν τρεις αναφορές ήδη από το 2010 και το 2011. Ήρθαμε σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές και ζητήσαμε πληροφορίες για το σχέδιο αυτό. Μας δόθηκαν λεπτομερείς πληροφορίες από πλευράς των Ρουμανικών Αρχών. Εξετάζοντας τις πληροφορίες αυτές στις 16 Δεκεμβρίου του 2011 ήδη, δύο χρόνια δηλαδή ακριβώς, στείλαμε τις πρώτες παρατηρήσεις μας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το γενικό συμπέρασμα σε εκείνη τη φάση ήταν ότι δεν είχε υπάρξει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, ε, κυρίως γιατί δεν είχε ακόμα δοθεί η άδεια εκμετάλλευσης. Η κατάσταση ηρέμησε για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι τον Αύγουστο του 2013 Εκεί η ρουμανική κυβέρνηση ψήφισε μια πρόταση νόμου, κατέθεσε μάλλον μια πρόταση νόμου, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαδικασία αξιολόγησης και θα μπορούσε επίσης να ε, επηρεάσει αρνητικά ε, τις κήτες των ποταμών της περιοχής. Λάβαμε πάρα πολλές επιστολές από πολίτες, από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και γι' αυτό παρενέβημε για μια ακόμη φορά και ζητήσαμε από τις Ρωμανικές Αρχές να μας δώσουν την πρόταση νόμου και την συμφωνία με την επιχείρηση εκμετάλλευσης χρυσού της Ρώσια Μοντάνα. Μας δόθηκε λοιπόν, οι πληροφορίες οι πρώτες μας δόθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου και το Νοέμβριο, τέλος Νοεμβρίου ζητήσαμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την εκτροπή των ποταμών. Οι Ρουμανικές αρχές δεν έχουν ακόμα απαντήσει, πάντως εμείς περιμένουμε μία απάντηση από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως την προηγούμενη εβδομάδα και η μέρα τρίτη αυτός, αυτή η πρόταση νόμου που δεν είχε ακόμα ψηφιστεί από τη Βουλή ε, μπήκε σε ψηφοφορία και απερίφθη. Η Επιτροπή λοιπόν παρακολουθεί την διαδικασία αδειοδότησης της μεταλλευτικής αυτής δραστηριότητας εμείς έχουμε σαν βασικό στόχο την πλήρη εφαρμογή των νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κανόνων και σε σχέση με τις εξορρυκτικές δραστηριότητες. Ουδεμία τέτοια δραστηριότητα δεν μπορεί να αναλυφθεί εκτός και αν υπάρχει πλήρης αδειοδότηση που να σέβεται την κοινοτική νομοθεσία ε, και τις οδηγίες ε, για την ε, εκ των προτέρων μελέτη των συνεπειών της δραστηριότητας αυτής και της εκμετάλλευσης των αποβλήτων κτλ. Εμείς πριν δύο χρόνια είχαμε πει βέβαια ότι μέχρι εκείνο το σημείο δεν είχαμε εντοπίσει κάποια παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας γιατί δεν υπήρχε ακόμα άδεια εκμετάλλευσης και η διαδικασία η εσωτερική αδειοδότησης συνεχίζεται και σήμερα είναι η ίδια ε, η, απάντησή μας. Ο κύριος Μποστινάρου. Επιτρέψτε μου να μιλήσω στα ρουμανικά για να χαιρετήσω εκείνους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Απευθύνω λοιπόν σε εσά ε, και σε όλα σε όλες τις χιλιάδες Ρουμάνων που παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή τη ε, μετάδοση και θέλω να τους πω το εξή. Πρώτον, εγώ δεν έχω επουδενή αλλάξει άποψη όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα και δεύτερον, προφανώς και παραμένω αντίθετος με την υλοποίηση αυτή του έργου. Επίσης, συμφωνώ ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Όχι να κλείσει όπως προτάθηκε σήμερα. Εγώ με κατά του κλεισίματος της ε, αναφοράς. Θέλω η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή, διότι πρέπει να εγγυηθούμε ότι η υλοποίηση αυτού του προγράμματος ε, θα γίνει με την ε, χρησιμοποίηση της ε, τελευταίας τεχνολογίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αναφέροντα από την Ένωση Αντάστρα για την ενημέρωση που μας έκανε και να πω ότι όταν πρότεινα να αναβληθεί η συζήτηση, κατ' ουσίαν είχα την άποψη που σας ανέφερα. Λυπάμαι που ο συνάδελφος δεν είναι ενημερωμένος τι ε, συνέβη στη Ρουμανία τις τελευταίες ημέρες. Ε, συστήθηκε μια ειδική των πραγμάτων επιτροπή που κατέληξε ότι θα πρέπει το πρόγραμμα να απορριφθεί. Το Κοινοβούλιο ομόφωνα ψήφισε υπέρ της ε, απόρριψης του αρχικού προγράμματος που είχε διαμορφωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Την ε, Τρίτη προχθές ε, το Κοινοβούλιο στη Ρωμανία λόγω των διαμαρτυριών, γιατί στη Ρουμανία υπάρχει τεράστια αντίδραση ε, απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα. Η κυβέρνηση λοιπόν της Ρουμανίας ξεκίνησε την εφαρμογή ενός άλλου προγράμματος που προβλέπει δύο καινοτομίες για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το ένα, το πρόγραμμα που βλάπτει το περιβάλλον, ζημιώνει το περιβάλλον αυτό σαφώς και απορρίπτεται και δεύτερον κανένας επενδυτής δεν θα μπορεί να εφαρμόζει τέτοιου είδους προγράμματα αν δεν χρησιμοποιεί και την τελευταία τεχνολογία. Εγώ λοιπόν ως Ρουμάνος και ως ε, περιβαλλοντολόγος ε, είμαι υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω αυτές οι προτάσεις δεν έγιναν αποδεκτές. Και συνέβη και το εξή. Η Επιτροπή πολύ σωστά μας λέει ότι ακόμα δεν έχει φτάσει η Επιτροπή Περιβαλλοντικού Αντικτύπου. Διότι το πρόγραμμα ακόμα δεν έχει εγκριθεί. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την έκκληση να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί περιβαλλοντικού αντικτύπου, δηλαδή την έκθεση Ζανόνη, που επιτρέπει να ε, εισαχθούν όλες αυτές οι δικές μας τροπολογίες, δηλαδή διαφάνεια, συμμετοχή της κοινωνίας των πελιτών, της κοινωνίας των πελιτών, ευθύνη των επενδυτών και πάρα πολλά άλλα συναφή. Αυτά τα στοιχεία δεν τα έχουμε από πλευράς Επιτροπής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε κατά νου ότι καλούμεθα να, τάσου, να δράσουμε ταχύτατα καθότι ολοκληρώνεται αυτός ο νομοθετικός κύκλος. Ο αναφέρον έρχεται από την Αγγλία, προέρχεται από την Αγγλία και πρέπει να πει σε όλους αυτούς τους ε, Ρουμάνους και εκείνους και εγώ ότι εδώ ε, συζητάμε για ένα επιχείρημα όπου δεν έχουμε όμως συγκεκριμένα στοιχεία. Θα ήθελα λοιπόν αυτή η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή, αυτό το υπογραμμίζω και θέλω να συζητήσουμε όταν θα έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες με βάση τις οποίες θα μπορούμε να απευθυνθούμε στον αναφέροντα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, υπογραμμίσουμε ότι όλα τα προγράμματα τα μελλοντικά στην ε, Ρουμανία ε, θα απαιτήσουν και την εφαρμογή των τελευταίων περιβαλλοντικών προδιαγραφών έτσι ώστε η Ρουμανία να μην γίνει κακό παράδειγμα για άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ουγγαρία που θέλουν να ξεκινήσουν την εξόριξη ορυκτού πλούτου. Εφόσον γίνεται κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο και γι' αυτό ευχαριστώ για άλλη μια φορά το αναφέρονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρο. Ο κύριος Χέλμερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι κάτι που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι το θέμα της Ρώσια Μοντάνα έχει γίνει στην ουσία ένα είδος ε, ποδοσφαίρου ε, σε πολιτικό επίπεδο και οι Ρουμάνοι πολιτικοί επιδιώκουν κάθε φορά τους εκλογικούς τους στόχους χτυπώντας τους αντιπάλους γύρω από το θέμα αυτό. Παρατήρησα ότι οι αντιρρήσεις από πλευράς του αναφέροντος είναι γενικού τύπου και θα μπορούσαν να ισχύσουν στις εξορρικτικές ε, δραστηριότητες και για χρυσό και για οτιδήποτε άλλο ε, αναπτυξιακή διαδικασία σε όλες τις χώρες. Και όταν τίθενται θέματα συγκεκριμένα όπως αρχαιολογικά ευρήματα και ε, προβλήματα σεισμικά ε, στην ουσία φαίνεται ότι είναι επιχειρήματα επιτούτου τα οποία χρησιμοποιούνται χωρίς να μας βοηθούν να καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση. Uh, λοιπόν, η Επιτροπή μας υπάρχει έτσι ώστε ε, να ε, συγκεντρώνεται η προσοχή μας σε θέματα παραβίασης του κοινοτικού νόμου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε μια μετρημένη απόφαση μέσα στην οποία μας είπαν ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν τα εξέτασαν. Το θέμα έχει προχωρήσει αρκετά, άδειε δεν έχουν δοθεί ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα δεν είναι σε θέση να μας πει ότι υπάρχει πιθανή παραβίαση του κοινοτικού νόμου. Δεν υπάρχει μάλλον παραβίαση του κοινοτικού νόμου. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να συζητάμε την αναφορά. Ε, η αλήθεια είναι ότι οι εξορρυκτικές διαδικασίες καλύπτονται από τις ρουμανικές νομικές ε, ρυθμίσεις και μιας και η Ρουμανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζονται και από τον κοινοτικό γενικότερα νόμο. Εγώ δεν είμαι και πολύ υπέρ του κοινοτικού νόμου όπως ξέρετε, αλλά τέτοιου είδους κανονισμού νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή, προσεκτική και εφαρμόζονται σωστά κάτω από συνθήκες τις οποίες υπάρχει υψηλό επίπεδο ανησυχίας του κοινού. Και εγώ ανησυχώ επίσης και για την προκλητική και καταχρηστική αντιμετώπιση της αρχής της πρόληψης. Γενικά ό,τι και να κάνουμε επικίνδυνο είναι. Όταν κατεβαίνουμε από το κρεβάτι μας το πρωί είναι πολύ επικίνδυνο. Όταν ανεβαίνουμε τα σκαλιά είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Γι' αυτό λοιπόν κάθε φορά κάποιοι βρίσκουν άλοθη για να μην κάνουμε ποτέ τίποτα. Υπάρχει όμως εδώ ένα ευρύτερο θέμα για το οποίο πράγματι ανησυχώ. Απαιτούνται επενδύσεις, απαιτείται ανάπτυξη, απαιτούνται θέσεις απασχόλησης, απαιτείται βιομηχανική δραστηριότητα. Και να μου επιτρέψετε να πω ότι η Ρουμανία είναι μια από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ανάγκη από βιομηχανικές δραστηριότητες περισσότερο από άλλους. Και αυτές οι πολύ μέτριες αντιρρήσεις που ακούστηκαν πρέπει να μας ανησυχούν γιατί τέτοιου είδους αντιλήψεις μπορεί να ισχύουν και σε άλλες χώρες. Έχω παραδείγματα και στη δική μου χώρα με μια αυτόματη αλλεργία σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια. Και έτσι βλάπτουμε τις επενδύσεις, βλάπτουμε το οικονομικό μέλλον, μέλλον της χώρας μας. Νομίζω λοιπόν ότι ο ρουμανικός λαός θα πρέπει να δει τα πλεονεκτήματα της πρότασης για τις δραστηριότητες αυτές του χρυσορυχείου και <clears throat> θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτές οι καθυστερήσεις μπορεί να οδηγήσουν τον επενδυτή στο να αποσυρθεί, να παρετηθεί και αυτό θα είναι εις βάρος του ρουμανικού λαού, εις βάρος της ρουμανικής οικονομίας εάν πράγματι φύγει ο, ομιλη, ο, επενδυτής από τη χώρα αυτή. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν που ε, άργησα να έρθω εδώ και αν όμως το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη αναφορά δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί δεν υπάρχει καμία παραβίαση του κοινοτικού νόμου. Πρέπει να κλείσει η αναφορά, είναι το πιο λογικό. Thank you, Mr. Elmer. Mrs. Κυρία Χάουκεν, από τους πιο θαραλέους συναδέλφους ο προλαλής σας. Δεν τον ενδιαφέρει αν δημιουργήσει εχθρούς. Οι περισσότεροι από μας αν είμαστε οι δύο γονείς Don't have any principle if is at stake. Uh, Θέλουμε να υπάρχει φρόνηση. Γι' αυτό ας παραμείνει ανοιχτή. Ίσως αυτή τη φορά να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε πρόληψη αντί εκ των υστέρων να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για λάθος. Χαίρομαι γιατί αυτή τη στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε εκ των προτέρων όλες τις πιθανές παραβιάσεις. Έχουμε και από άλλες χώρες αναφορές, Βουλγαρία, Ελλάδα και ξέρω ότι όλοι μας παρακολουθούν, μας προσέχουν και πρέπει όλα αυτά να μπορούμε να τα λαμβάνουμε υπόψη μας πριν γίνει κάποιο ατύχημα. Η αντίδραση στην Ρουμανική Βουλή σε τέτοιου είδου ανησυχίες βασίζεται. Αλλά πέστε μου εσείς, εάν είναι βέβαιο ότι στη νέα νομοθεσία θα λαμβάνεται υπόψη αυτό το θέμα της πρόληψης, γιατί επανειλημμένως πάρα πολλές φορές έχουμε περιοριστεί στη διαπίστωση εκ των υστέρων. Συνήθως όταν υπάρχουν υψηλά κέρδη σημειώνονται και πολλές παρανομίες. Καταρχήν λοιπόν ευχαριστώ την Κομισιόν για την καλή της απάντηση. Το Ρουμανική Βουλή γιατί έκανε τον κόπο να εφαρμόσει κάποια φρόνηση και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για το ότι μπορούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις πριν γίνει το κακό και θα ζητούσα από τους πολίτες της Ρουμανίας και των άλλων χωρών να συνεχίσουν να προσέχουν τέτοια θέματα και να μας πληροφορούν γιατί δεν νομίζω ότι ο χρυσός είναι από τα πιο απαραίτητα αγαθά στον κόσμο. Μπορώ να φανταστώ άλλα σχέδια και προγράμματα που να φορούν πολύ πιο απαραίτητα προϊόντα και να δημιουργούν και περισσότερες θέσεις απασχόλησης αντί, αυτά τα, αντί για αυτά τα χρυσορυχεία. Βέβαια δεν είναι δικό μας θέμα. να τα βλέπουμε όλα αυτά, αλλά αν είναι αλήθεια αυτά που έχω μάθει, Πρέπει να το προσέξουμε. Να το κρατήσουμε ανοιχτό λοιπόν και ελπίζω και η Κομισιόν να το παρακολουθεί. έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα θα γίνουν όπως πρέπει με το σωστό EEA δηλαδή. Ο κύριος Αγκουράκης.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 Πρέπει, επαναλαμβάνω, να παραμείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη αναφορά. Αυτό για ποιο λόγο. Πρώτον γιατί θεωρώ αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας το οποίο έχει οργανωθεί στην Ρουμανία έχει πάρα πολύ μεγάλη λαϊκή βάση για έναν απλό λόγο, γιατί οι διαμαρτυρόμενοι έχουν δίκιο. Δεν υπάρχει καμιά άλλη εξήγηση σε αυτό, δεν πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε άλλους λόγους για τους οποίους έχει διαμορφωθεί ένα τόσο ισχυρό κίνημα. Και τώρα εδώ να έρθω σε κάτι το οποίο έχει ήδη αναφερθεί. Γνωρίζετε ότι δυστυχώς η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι συνήθως καθυστερημένη χρονικά Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί δεν υπήρχε τελική απόφαση γύρω από το συγκεκριμένο αυτό σχέδιο. Ε, συνήθως όταν έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει οτιδήποτε για να τις ακυρώσει αν για κάποιο λόγο βρει ότι δεν τις κάνουν. Τρίτον, η απόφαση της Ρωμανικής Βουλής. Νομίζω ότι ε, χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλά επιχειρήματα, τεχνικά επιχειρήματα, κοινωνικά, οικονομικά, τα οποία οδήγησαν την Ρουμανική Βουλή στη συγκεκριμένη απόφαση. Υπάρχει και άλλο ένα επιχείρημα και θέλω να συνδέσω το επιχείρημα με αυτό, με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί και στην Ελλάδα έχουμε μια αντίστοιχη περίπτωση. Και στην Ελλάδα υπάρχει ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση για το περιβάλλον. Ε, αυτά τα οποία, για τα οποία φοβόμαστε, κανένας δεν μας δίνει εγγυήσεις ότι δεν θα συμβούν. Συνεπώς οι λαϊκές αντιδράσεις είναι ισχυρότατες. Λυπάμαι λοιπόν που άκουσα <coughs> να κάποιες απόψεις σε αυτήν εδώ την αίθουσα που λέγουν ότι η δημιουργία ενός τοπίου ε, περίπου σεληνιακού γιατί για κάτι τέτοιο μιλάμε έτσι μετά την εξορρυκτική δραστηριότητα ένα τέτοιο τοπίο θα δημιουργηθεί ε, κάποιοι πιστεύουν ότι ένα τέτοιο τοπίο θα βοηθήσει στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της Ρωμανίας. Ε, τώρα αυτό ε, είναι μια αντίληψη την οποία θα χαρακτήριζα νεοαπικιακή. Ε, δεν είναι κάτι που έχει ανάγκη η Ρουμανία αυτή η οικονομική δραστηριότητα. Ούτε η Ελλάδα έχει ανάγκη ε, μια τέτοια οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη. Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή. Κρατήστε παρακαλώ τη συγκεκριμένη αναφορά ανοιχτή έχουν ακουστεί πάρα πολλά επιχειρήματα τα οποία συνδέονται με το μέλλον της χώρας. Ας μην μιλάμε μόνο για το παρελθόν, ας μην μιλάμε πράγματι μόνο για τα αρχαιολογικά ερήπια, ας μην μιλάμε μόνο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ας μιλήσουμε για το πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης. Έχει το λόγο αναφέρον ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την απάντησή της, απαντώντας την απάντησή της και στις παρατηρήσεις του κυρίου Χέλμερ να επαναλάβω κάτι το οποίο είπα. Εμείς επικαλούμεθα την αρχή της πρόληψης για έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Δεν ζητάμε την αρχή της, ε, την, ε, την εφαρμογή αυτής της αρχής για, γενικά γνωρίζουμε τι θα συμβεί αν τυχόν η δραστηριότητα αυτή αδειοδοτηθεί. Γνωρίζουμε ότι μία περιοχή την οποία χιλιάδες αρχαιολόγοι και ιστορικοί αναγνωρίζουν σαν πολύ μεγάλη σημασία μετατραπεί σε ένα λατομείο. Και γι' αυτό ακριβώς ζητάμε την, αρχή της, την εφαρμογή της αρχής της πρόληψης, γιατί γνωρίζουμε τι θα ακολουθήσει αν λειτουργήσει το σχέδιο γνωρίζουμε από τώρα. Είναι σαφές το τι θα ακολουθήσει. Σας, Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν η αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή διότι η πλειοψηφία αυτό ζήτησε. Αλλά μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο κύριος Έλμερ. Θέλω να τονίσω ότι εμείς φροντίζουμε πάντοτε να κάνουμε κάτι για να προλάβουμε για την πρόληψη όχι μόνο για να υποστηρίξουμε τη δημιουργία και λειτουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορεί παρά μόνο να παρέμβει κατόπιν εορτής. Αυτή είναι η δουλειά μας και το αναγνωρίζουμε αυτό. Αυτό είναι ο, ο αναγνωρισμένος στόχος μας. Αυτό προσπαθούμε κάθε φορά που εργαζόμαστε εδώ. Αλλά δεν το καταφέρνουμε βέβαια. Και πάντοτε υπάρχει κομισιόν που μας λέει ότι δεν μπορεί να παρέμβει διότι δεν έχει ακόμα υπάρξει παραβίαση. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Θα παραμείνει ανοιχτή και θα περιμένουμε περαιτέρω επεξεργασία από την Κομισιόν. Τώρα το επόμενο θέμα που είναι αναφορά από την Γαλλική Ένωση Άριβεμ για την κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής φυσικού αερίου στην Ρομενβίλ. Μαζί με μια άλλη παρόμοια αναφορά άλλου Γάλλου πολίτη για την προβλεπόμενη θέση εργοστασίου μεθανιοποίησης πάλι στο Ρομενβίλ. Δεν είναι παρόντες οι αναφέροντες. Μπορώ όμως να δώσω το λόγο αμέσως στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Ντέιβιτ Γκριμό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Χαίρετε. Θα σας μιλήσω για την αναφορά αυτή. Να σας πω σύντομα τα γεγονότα. η οργή των αναφερομένων και οι πρωτοβουλίες της Κομισιόν ως αντίδραση. Λοιπόν, γιατί πρόκειται, πρόκειται. Είναι ένα σχέδιο εκμετάλλευσης μιας παραγωγής μιας μονάδας ε, διαχείρισης των αποβλήτων κοντά στο Παρίσι, η οποία συνήθως ονομάζεται μεθανιοποίηση καθώς και ένα κέντρο ε, διαχείρισης ε, ογκωδών αντικειμένων. Έχει χαρακτηριστεί γενικού συμφέροντος ή ενδιαφέροντος έργο γιατί θα εξυπηρετεί 22 κοινότητες εκτός Παρισίων και δύο περιφερειών του Παρισιού. Οι αναφέροντες μιλούν για ενοχλήσεις που δημιουργεί εκπομπή ρήπων και η οσμή, δυσάρεστη οσμή. πρέπει να ξέρετε ότι έτσι όπως υποβλήθηκε η αναφορά μιλούσε γενικά, δεν είχε νομικά επιχειρήματα ιδιαίτερα ή συγκεκριμένα. Λοιπόν, ημερομηνίε. Η αίτηση αδειοδότησης υποβλήθηκε από την εταιρεία τον Μάιο του 2009. και η νομαρχιακή άδεια χορηγήθηκε στην εταιρεία τον Ιανουάριο του 11. Μετά όμως δεν άρχισαν αμέσως οι εργασίες και μάλιστα σταμάτησαν γιατί, γιατί κηρύχθηκε μορατόριο από την 1η Φεβρουαρίου 2012 για να εξεταστούν τα αιτήματα των περιοίκων, μεταξύ των οποίων και οι αναφέροντες. Για επανεξέταση λοιπόν του προγράμματος. Το μορατόριο ισχύει ακόμη. Έχουν γίνει έλεγχοι δύο από το ΙΝΕΡΙΣ και από το ΡΕΠ δύο γαλλικά Ινστιτούτα για περιβαλλοντολογικά θέματα που κατέληξαν ότι οι μελέτες περιβαλλοντολογικής αξιολόγησης είχαν γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εθνική νομοθεσία και έκαναν και ορισμένες συστάσεις. Τα συμπεράσματα των ελέγχων είναι δημόσια και συζητήθηκαν και δημόσια. Η εταιρεία και ιδιαίτερα το Συμβούλιο των Ενδιαφερομένων ε, Κοινοτήτων αποφάσισε να δεχτεί όλα τα συμπεράσματα των δύο εθνικών αυτών Ινστιτούτων Ελέγχου. Αναθεώρηση λοιπόν των όρων της αδείας που είχε δοθεί. Τι έκανε η Κομισιόν λοιπόν. Υπάρχουν δύο γραπτές δηλώσεις από τον Νοέμβριο του 12 και τον Φεβρουάριο του 13 που στάλθηκαν στην Επιτροπή σας και μία τρίτη γραπτή ανακοίνωση ή δήλωση που υποβλήθηκε πιο πρόσφατα πριν από μερικές μέρες σε εσά πάλι. Η Κομισιόν άρχισε, άνοιξε ένα φάκελο EU Pilot που λέμε που επιτρέπει στην Κομισιόν να θέσει επισήμως ερωτήματα στις γαλλικές αρχές για το πρόγραμμα. Οι γαλλικές αρχές απάντησαν το καλοκαίρι του 2013 και επιβεβαίωσαν τα εξής. Οι συστάσεις των δύο Ινστιτούτων πράγματι θα εφαρμοστούν. Τι λένε οι συστάσεις. Να σας πω δύο-τρεις από αυτές. Βελτίωση της ασφαλείας του εργοστασίου εγγύηση ενισχυμένων ελέγχων και εγγύηση της ε, ικανοποίησης των παραπώνων για ενόχληση από την κακοσμία. Με βάση λοιπόν την απάντηση αυτή των γαλλικών αρχών, η Κομισιόν έκρινε τα εξής το σχέδιο δεν καλύπτει την οδηγία IPPC, αλλά την νέα οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές. Πρέπει να, έπρεπε να δούμε λοιπόν αν συμφωνεί με αυτήν την οδηγία του 2010. Δεύτερον, το σχέδιο δεν καλύπτεται από τη γενικότερη νομολοθεσία για τις περιβαλλοντολογικές αξιολογήσεις γιατί έγινε εθνικά. Τρίτον, το σχέδιο δεν αφορά την οδηγία σε Βέζο 2 γιατί έχει πολύ μικρό όγκο επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων. Δεν είναι τοξικά τα απόβλητα που θα χρησιμοποιεί, που θα διαχειρίζεται. Και τέλος, πληροφορηθήκαμε ότι έχουν γίνει και νομικές προσφυγές ενώπιον του αρμόδιου γαλλικού δικαστηρίου. Μία από αυτές την υπέβαλε ένας από τους αναφέροντες. Το Διοικητικό Δικαστήριο του Μοντρόιγ, στα περίχωρα του Παρισιού, εξέδωσε απόφαση τον Απρίλιο του 2013 και η απόφαση αυτή ακυρώνει την άδεια που είχε χορηγηθεί, την άδεια εκμετάλλευση διότι λέει είχε κενά η περιβαλλοντολογική μελέτη αξιολόγηση. Έγινε όμως ε, έφεση προς το ίδιο διοικητικό δικαστήριο και θα αποφανθεί στις 16 Ιουνίου του 2014. Τι θα γίνει τώρα λοιπόν. Αν το διοικητικό εφετείο επικυρώσει την απόφαση του προηγουμένου δικαστηρίου πρέπει η εταιρεία τότε να καταθέσει νέο πρόγραμμα και να αρχίσει ολόκληρη νέα διαδικασία. Αν όμως το εφετείο, το διοικητικό εφετείο δικαιώσει την εταιρεία, τότε οι γαλλικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα τροποποιηθεί η άδεια που είχε χορηγηθεί για να συμφωνεί με τις συστάσεις των δύο Ινστιτούτων. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ο Πέτρος Γιάρ. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι η Κομισιόν εξήγησε με πολύ εντυπωσιακό τρόπο ότι η όλη διαδικασία βρίσκεται, εξελίσσεται. Ακόμα η δεν έχει ληφθεί η δικαστική απόφαση, δεν έχει αποφανθεί το δικαστήριο. Από την άλλη οι γαλλικές αρχές και αυτές δεν έχουν δραστηριοποιηθεί. Εγώ θα έλεγα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και παρακαλούμε την ε, Κομισιόν να μας ενημερώσει αν προκύψει κάτι καινούριο. Ε, Παραδείγματος χάρη ε, όταν ε, θα έχει εκδοθεί απόφαση, τότε μπορούμε ίσως ε, να ξαναδούμε την όλη υπόθεση. Εγώ είμαι αρκετά ενημερωμένο για όλη αυτή την υπόθεση, γιατί και εσείς υπενηχθήκατε ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ήδη γίνονται κάποιες βελτιώσεις που ικανοποιούν τον αναφέροντα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Αυτό είναι κάτι που το κρατάω στα συν. παρακαλώ όμως η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή. Κυρία Χόκαν, κυρία θέλω να πω ότι δεν μου αρέσει που αυτό το έγγραφο το έχουμε μόνο στα γαλλικά, γι' αυτό εγώ δεν θα συμμετέχω. Αλλά εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό όμως. Okay, thank you. Nobody else. Άλλος παρακαλώ, επιθυμεί κάποιος άνος το λόγο, από ό,τι βλέπω όχι, κατόπιν τούτου Παραμένει ανοιχτή αυτή η αναφορά, όπως το ζητήσατε, κλείνει η συζήτηση και πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι η ψηφοφορία. Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη στη Γαλλικία. Η κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πέντε λεπτά. Στις έξι ώρα ψηφίζουμε. Λοιπόν, Δεν μπορείτε να παραβιάσετε ε, το δικαίωμά μας να έχουμε συζήτηση πριν από την ψηφοφορία. Σας παρακαλώ κύριε Χόκερ, μισό λεπτό. Εγώ είπα ότι στις 6 ώρα θα γίνει η ψηφοφορία για να μπορούν να έρθουν τα μέλη. Και τώρα λοιπόν δίνω το λόγο στην κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, ε, έχω ένα ερώτημα. Ε, στις 12 και 4 ο πρόεδρος Σούλτς ε, σας έστειλε ένα email και θέλω να ρωτήσω κατά πόσον παρόλα αυτά θα ψηφίσουμε ή μήπως λαμβάνοντας υπόψη αυτά που είπαν οι Στάλτη Στανούκο και εγώ ήδη την τελευταία φορά, μήπως ε, προτίθεστε να αναβάλλετε την ψηφοφορία. Uh, did Σας κατάλαβα. Περίμενα να τελειώσετε την παρουσίασή σας, την παρέμβασή σας. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση, λέει η κυρία Τφέρτμαν. Στην περίπτωση που δεν αναβληθεί τώρα η ψηφοφορία, η Τατιάνα Σδάνοκα και εγώ καταθέσαμε τροπολογίες στις συστάσεις όταν ε, δεν γνωρίζαμε ακόμα ότι το περιγραφικό κομμάτι ε, θα είχε αλλάξει επί της ουσίας, ε, τότε είχαμε καταθέσει τις τροπολογίες. Πέραν αυτού, η διαφοροποιημένη άποψη την οποία προετοιμάσαμε εγώ και η Τατιάνα θα πρέπει να προσαρτηθεί παρακαλώ στο κείμενο εργασίας και να γίνει και αυτό σαν τέτοια άποψη διαφορετική δεκτή από την Επιτροπή. κυρία Σντάνοκα. Yes. Ήδη έχω εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν πήρα μέρος στην συζήτηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης, γιατί τα έγγραφα τα οποία κατετέθησαν προς ψηφοφορία σήμερα Νομίζω ότι είναι καρπός παραβίασης των κανόνων. και δεν γίνεται σεβαστός, το, δεν γίνεται σεβαστό το συγκεκριμένο άρθρο το οποίο έχει επικυρώσει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεπώς λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε μέρος στην ψηφοφορία σήμερα γιατί παρότι έχουμε καταθέσει τροπολογίες όπως ε, είπε ήδη η Αγγέλικα Βέρτμαν όταν καταθέσαμε τις τροπολογίες δεν γνωρίζαμε ότι το περιγραφικό τμήμα ε, θα άλλαζε βασικά και το οποίο είχε προταθεί χωρίς διαβούλευση και χωρίς καμία δυνατότητα αλλαγής. Παρά την πλειοψηφία η οποία είχε διαμορφωθεί στο εσωτερικό της αντιπροσωπείας των τριών. Κανονικά ε, η άποψη, η αποκλίνουσα άποψη είναι άποψη της μειοψηφία, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι μία μοναδική περίπτωση στη δημοκρατία όπου η άποψη της πλειοψηφία είναι η αποκλίνουσα άποψη. Έτσι λοιπόν εμείς ε, δεν θα συμμετέχουμε στη ψηφοφορία. Η κυρία Χόκεν. Κοιτάξτε, έχω σοκαριστεί φοβερά. Έχουμε εδώ κανόνες, σαφείς, και βλέπουμε ότι επανειλημμένος παρόλα αυτά δεν μας προστατεύουν οι κανόνες. Ακόμη και αν μία πλειοψηφία δηλαδή θέλει να συνεχίσει να παραβιάζει τους κανόνες, το κάνει. Δεν είναι σωστό. I think it's undermining uh, our... Και λυπάμαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Η θέση της Αγγελικής και της κυρίας Δανόκα είναι ότι πρέπει όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν. Αν δεν είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε όλοι, τότε μπορούμε και να σταματήσουμε τελείως. Ευχαριστώ λοιπόν. Εκφράσατε τις θέσεις σας και η μεν και η δε. Έχουμε τα έγγραφα και ευχαριστώ την κυρία Σδανόκα και την κυρία Βέρτμεν που έκαναν τον κόπο να γράψουν επιστολή στον κύριο Σούλτς και στον κύριο Σούλτς που μου έστειλε απαντητική επιστολή όπου υποστηρίζει την απόφασή μου. Μια στιγμή κυρία Σδανόκα, μια στιγμή είναι δημόσιο έγγραφο η επιστολή αυτή και λέει Είμαι, λέει ο κύριος Σούλτς, είμαι βέβαιος ότι στο ρόλο σας ως Προέδρου της Επιτροπής σας θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να επέλθει κάποια συνένεση σύμφωνα με τον κανονισμό. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε παραπάνω. Και αυτή είναι η ερμηνεία μου του κανονισμού στην οποία κατέληξα διαβάζοντας γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και της ΑΦΚΟ. Νομίζω λοιπόν ότι κάνω αυτό που μου ζήτησε να κάνω ο πρόεδρος Σούλτ. Τώρα λοιπόν είμαστε στην ψηφοφορία και δεν μπορούμε να συνεχίζουμε συζητήσεις. Αρχίζει η ψηφοφορία και όπως μου ζήτησε γραπτός ο κύριος Σούλτς θα τον πληροφορήσω στη συνέχεια για τα αποτελέσματα. λάβω την ευθύνη της εκτέλεσης της απόφασης που έλαβα όσο αμφιλεγόμενη και να είναι η κατάσταση. Λοιπόν αυτή είναι η ευθύνη μου, αρχίζει η ψηφοφορία. Πώς τι... Σας παρακαλώ κυρία Χάουκεν μου. Ορίστε εσείς τελευταίος για διαδικαστικό. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε η κυρία Στάνοκα γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι σε αυτήν την έκθεση παρά μόνο η έκφραση της άποψης της μειοψηφίας. Κατανοώ βέβαια την θέση της κυρίας Ντάνοκα. Εγώ έχω την ευθύνη να ψηφίσω κανονικά, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο λειτουργεί εις βάρος ε, της ίδιας αξιοπιστίας του Κοινοβουλίου η διαδικασία που ακολουθήσαμε και θα πληρώσουμε τις συνέπειες. Thank you. Now I am opening the, the vote. Ωραία, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Λοιπόν, τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. αποχές ηλεκτρονική επανάληψη έληξε όχι έληξε έληξε Okay, but we have. Uh, okay, Είπα έληξε, αλλά θα την ξανακάνουμε την ψηφοφορία. Μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή. Να είπα μια στιγμή. Θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Πρέπει να σας πληροφορήσω καθώς και τον κύριο Γιάρ ότι μόνο 11 μέλη υπάρχουν και τώρα ψηφίζουν 13. Παρακαλώ λοιπόν κύριε Γιάρ, 11 μέλη σας ψηφίζουν. Yes, to Mr. Yar. So. So, two please. Δύο να απόσχουν παρακαλώ, να μην ψηφίσουν. 11 από το ΕΛΚ μόνο, κύριε Γιάρο. Έντεκα. Point of order. Point of order. No, no, we have to be 12. Όχι, 12 πρέπει να είμαστε, 12. Διαδικαστικό. Κοιτάξτε, διαδικαστικό επιμένω. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει 12 μέλη, Πρόεδρε, 12. Κάθε φορά ψηφίζουμε και τώρα μου λέτε ότι είμαστε 11. Όχι, 12 είναι οι ψήφοι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και γι' αυτό παρακαλώ ε, να το καταλάβει αυτό και η γραμματεία όταν λέει ότι είναι 11 είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και πρέπει να μας δώσει εξηγήσεις γιατί μας βγάζει 11. Ε, είναι σαν να παίρνει η γραμματεία μία ψήφο της πολιτικής μας ομάδας. On the point of order. Κυρία Φερνάντες διαδικαστικό και εσύ. Κύριε Φερνάντες. Ναι, ξέχασα την κάρτα μου στο Στρασβούργο. I will vote like that. Okay, thank Ωραία. Λοιπόν, και εγώ διαδικαστικό κύριε Χάουκεν. Όχι μια στιγμή, σας παρακαλώ. Όλοι όσοι θα ψηφίσουν έχουν γραφτεί από την αρχή, όχι και οι αναπληρωματικοί. Όχι, όχι κυρία Χάουκεν, δεν είναι. πρέπει να είναι παρόντες όλοι όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου. Λοιπόν, 12 μέλη του ΕΛΚ διορθώνω και μόνο 12. Άρχεται πάλι η ψηφοφορία λοιπόν για τη δεύτερη τροπολογία. Άρχισε η ψηφοφορία. Έληξε. 13 υπέρ 10 κατά καμία αποχή. Α, 10 και 1 είναι 1. Ναι. Κατά και καμία αποχή. Η τροπολογία εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Α, είναι οι ίδιες, έως πάνω, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 σε 2 τμήματα. Το πρώτο τμήμα σε 2 τμήματα. Σε 2 τμήματα. Μα εδώ γράφει inadmissible. Εγώ την θεώρησα αποδεκτή admissible. Σε δύο όμως τμήματα. Το πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Μάλιστα. pour savoir, Madame la Présidente, puisque... Κοιτάξτε κυρία Πρόεδρε, η τροπολογία αυτή χωρίστηκε σε δύο τμήματα, αλλά πρέπει να ξέρουμε σε τι ακριβώς τμήματα. Εμείς το ΕΛΚ προτείνουμε να δεχτούμε το τμήμα το τμήμα που δεν αφισβητεί τα περί της Φερόλ ή Σερόλ. Παραμένει πάντως προς ψήφιση. Λοιπόν, το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 4 χωρίς τη λέξη Φερόλ. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα, αυτό είναι το πρώτο τμήμα, χωρίς φερόλ. Ποιος είναι υπέρ. Without the word Χωρίς τη λέξη φερόλ. Χωρίς. Τη λέξη φερόλ. Κατά. Κανείς. Αποχές. Το πρώτο τμήμα λοιπόν εγκρίθηκε ομόφωνα και πανψηφί. Άρα το δεύτερο μάλλον απορρίπτεται. Όχι, α, δεν, όχι απορρίπτεται, αλλά να, καταπίπτει κατά κάποιον τρόπο. Ώρα τροπολογία 6 τώρα, υπέρ κατά αποχές πρέπει να επαναλάβουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Να προσθέσουμε και τον κύριο που δεν έχει την κάρτα του. Λοιπόν, 12 υπέρ και εγώ ψήφισα λάθος, διορθώνω. 13 υπέρ με τον κύριο εδώ. 12 υπέρ, είπα, 12 υπέρ. Και 13 κατά με τον Κύριο. Έχει απορριφθεί η τροπολογία. Τροπολογία 7 με προφορική τροποποίηση. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροποποίησης? Όχι. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ της 7 με την προφορική τροποποίηση? Κατά. Πάλι επαλήθευση προτείνω όλο να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά γιατί αλλιώς είμαστε πολλοί λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία για την 7. Έληξε. 11 υπέρ 13 κατά καμία αποχή. Όχι, 11 και 1, 12 υπέρ. 12 υπέρ. Μα αυτό είπα 11 συν 1, 12 δηλαδή. 11 συν 1, 12. 12 υπέρ, 13 ψήφοι κατά καμία αποχή. Απορρίπτεται. Η 8 έχει αποσυρθεί αν εγκριθεί λέει η 7 μάλιστα. Τροπολογία 9. είναι ασαφής η διατύπωση. Λέει αποσύρεται εάν εγκριθεί η 7. Έτσι λέει. Η προφορική τροποποίηση είχε γίνει δεκτή αλλά η 7 με την προφορική είχε αποσυρθεί. Α, ναι, σωστά, σωστά. Τώρα λοιπόν, τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. 8. Έληξε. Ε, ωραία. Έληξε είπα. 11 συν 1 υπέρ, 13 κατά καμία αποχή. Απορρίπτεται. 9 άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. 6 υπέρ. Κύριε Φερνάντες, υπέρ. 6 ε, και 1, 7 υπέρ. 13 κατά 5 αποχές απορρίπτεται. Amendments. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Close the... Έληξε. Έληξε. 24 ψήφοι υπέρ, τίποτε άλλο, πανψηφί. 12 άρχεται η ψηφοφορία. 12 έληξε. Εγκρίνεται πανψηφί 23 υπέρ. 24 δηλαδή, 24. 13. Άρχεται. έληξε. Όχι, όχι, όχι. Α, ναι. Α, τότε καλά. Λοιπόν, πέντε υπέρ, είκοσι κατά, καμία αποχή. Ναι, καλά και, και ένας ακόμη υπέρ, έξι υπέρ. Απορρίπτεται. 14, τροπολογία 14, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχισε. Έληξε. 5 συν ένας υπέρ, 13 κατά, 6 αποχές. Απορρίπτεται. 15 άρχισε η ψηφοφορία. Έληξε. 13 υπέρ, 12 συν 1 κατά, πάλι 13, ισοψηφία, καμία αποχή απορρίπτεται. 16, 13 απορρίφθηκε η προηγούμενη απορρίφθηκε 13-13. Λοιπόν, τώρα η 16. 16. Άρχισε η ψηφοφορία ήδη. Έληξε. Πάλι 13-13. Α, υπέρ, δεν ψηφίσατε εσείς, υπέρ. 13 υπέρ, 13 υπέρ, 13 κατά, Απορρίπτεται. Όπω πριν. Λοιπόν, 17. Άρχεται η ψηφοφορία. 17. Μια στιγμή να το υπολογίσω. Θα ήθελα να ζητήσω από τη Γραμματεία να διευκολύνει τις ψηφοφορίες, εν πάση περιπτώσει. Παρακαλώ η Γραμματεία να διευκολύνει τις ψηφοφορίες. Τώρα λοιπόν τροπολογία 18 Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. 6 υπέρ, 5 και 1 δηλαδή, 11 κατά 8 αποχέ. Απορρίπτεται 19. Άρχεται. Έληξε. 13-13 πάλι. Δηλαδή 13 και 12 συν 1. Απορρίπτεται. 20. Έληξε. 5 συν 1 σε 6 υπέρ, 12 κατά 8 αποχές απορρίπτεται. 21 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Δώδεκα συν ένα με δεκατρία. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Έληξε. 5 και ένας 6, 13 κατά 7 αποχές απορρίπτεται. 22 άρχεται. Άρχισε. Έλξε. 6 υπέρ 20 κατά. Απορρίπτεται. 23 μα άρχεται. έληξε. Τέσσερις υπέρ υπέρα κατά δύο αποχές απορρίπτεται. 24 αρχίζει, άρχισε. Έληξε. Δώδεκα υπέρ 6 και 1 κατά 7 αποχές εγκρίνεται. 25 άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. 5 συν ένας υπέρ, 12 κατά 9 αποχές, απορρίπτεται. 26 άρχεται έληξε. «27 ομόφωνα υπέρ». Μερικοί δεν ψηφίζουν φαίνεται. 27 υπέρ, άρχεται η ψηφοφορία, 27 τροπολογία, άρχεται η 27 τροπολογια αρχεται έληξε. 24 υπέρ, μία αποχή. εγκρίνεται 28 άρχεται έληξε 5 και 1 υπέρ 12 κατά 9 αποχές απορρίπτεται 29 αρχίζει άρχισε έληξε 20 υπέρ, 3 και 1 κατά, δύο αποχές εγκρίνεται. 30 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα αρχίζει η ψηφοφορία. Έληξε. 27 ομόφωνα υπερ δεύτερο τμήμα. Άρχισε. Έληξε. 13-13. Απορρίπτεται. 31 άρχισε η ψηφοφορία. Έληξε. Έξι υπέρ 11 κατά, 9 αποχές. Απορρίπτεται. 32. Άρχισε, έληξε. 21 υπέρ, 5 και 1 κατά, εγκρίνεται. 33 έχει καταπέσει. 34 Αρχίζει η ψηφοφορία. Έληξε. Ψηφίζουν όλοι. Είπα έληξε. Πέντε και ένας υπέρ. 20 κατά απορρίπτεται. Μια στιγμή, συνάδελφοι. Yeah, there's only six, I suppose. Yes, it's okay. We are all serious, I hope. But Secretariat is very serious, so one... Η γραμματεία είναι πολύ σοβαρή και θέλει να επαληθεύσουμε. Και συμφωνώ και εγώ. Τροπολογίες, τροπολογία 35 πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Close the vote έληξε 26 υπέρ μία ψήφος κατά εγκρίνεται εγκρίνεται δεύτερο τμήμα άρχεται ψηφοφορία έληξε Κατά πίπτη 13-14. 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. 26 υπέρ, μία αποχή εγκρίνεται. 37 άρχεται. Έληξε. 27 ομόφωνα υπέρ εγκρίνεται. 38 άρχεται έληξε 26 υπέρ μία αποχή εγκρίνεται 39 άρχεται έληξε

απορρίπτεται. 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, έληξε. 6 υπέρ 11 κατά 9 αποχές απορρίπτεται. 42. Άρχεται. έληξε 6 υπέρ 12 κατά 9 αποχές απορρίπτεται 44 άρχεται έληξε 6 υπέρ 12 κατά 9 αποχές απορρίπτεται 43 άρχεται η ψηφοφορία έληξε 14 υπέρ, 13 κατά εγκρίνεται. 45 αρχίζουμε την ψηφοφορία, έληξε. Έληξε. 13, 14 δηλαδή υπέρ, 11 κατά εγκρίνεται. 46 άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. 6 υπέρ 12 κατά 8 αποχές απορρίπτεται. 47 άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. 5 υπέρ 12 κατά 9 αποχές απορρίπτεται. 48 Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. 6 υπέρ 13 κατά 8 αποχές απορρίπτεται. 49 άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. 26 υπέρ και μία αποχή. Εγκρίνεται. 50 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. 25 υπέρ, μία αποχή. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. 18 υπέρ 8 κατά μία αποχή εγκρίνεται. 51 άρχεται η ψηφοφορία. 13 υπέρ 6 κατά 8 αποχές εγκρίνεται. 52 άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. 6 υπέρ 20 κατά μία αποχή απορρίπτεται. 53 άρχεται. Έλήξε. 6 υπέρ 20 κατά μία αποχή απορρίπτεται. 54 αρχή. Τέλος. 21 υπέρ 6 κατά εγκρίνεται. 55 γιατί έληξε. Έξι υπέρ 20 κατά απορρίπτεται. 56 αρχή. Τέλος. 20 υπέρ 6 κατά εγκρίνεται. 57 αρχή. Τέλος. Έξι υπέρ 12 κατά 9 αποχές απορρίπτεται. 58 αρχή. Έλος. 13 υπέρ 12 κατά μία αποχή εγκρίνεται. 60 αρχή. Τέλος. Έξι υπέρ 21 κατά απορρίπτεται. 61 αρχή. Τέλος. 6 υπέρ 13 κατά 8 αποχές απορρίπτεται. 62 αρχή. Ε, τέλος. 6 υπέρ 21 κατά απορρίπτεται. 63. Έχει καταπέσει, έχει καταπέσει. Α, όχι, δεν έχει καταπέσει. 63 έλξε. «22 υπέρ και 4 αποχές». Εγκρίνεται. 64. Και 65. Είναι ταυτόσιμες για διαγραφή, για διαγραφή, για διαγραφή. Διαγραφή. Η 64 είναι ίδια με την 65 ή το ανάποδο. So we can vote together six... Μαζί 64 και 65. Αρχη, Τέλος. Τέλος είπα. 12 υπέρ, κύριε Φερνάντε, στη... Α, 13 υπέρ, 13 κατά. Εσείς τι είπατε, υπέρ και εσείς. Α, 14 υπέρ τότε και 13 κατά, εγκρίνεται. Είμαστε 27 με τον κύριο Φερνάντες που δεν έχει κάρτα. Δεν έχει κάρτα. Ελέγξαμε τους αριθμούς σοσιαλιστών και ΕΛΚ και είναι εντάξει οι αριθμοί είναι. 66 άρχεται η ψηφοφορία έληξε 26 υπέρ εγκρίνεται. 67 άρχεται η ψηφοφορία. Έλξε. 20 υπέρ 6 κατά εγκρίνεται. 68 άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. 21 υπέρ 6 κατά εγκρίνεται. 69 άρχεται η ψηφοφορία, έληξε. 2 υπέρ 16 λέει η πρόεδρο, κατά 8 αποχές απορρίπτεται, 70 άρχεται, έληξε. 17 υπέρ μία ψήφο ε, κατά 8 αποχές εγκρίνεται. Ε, εγκρίνεται, εγκρίνεται. 71. Άρχεται. Έλξε. 14 υπέρ, 13 κατά, εγκρίνεται. 72 άρχεται. Έλξε. 14 υπέρ, 13 κατά. Εγκρίνεται. 73 αρχή. Τέρμα. 15 υπέρ, 11 κατά. Εγκρίνεται. 74 αρχή. Αρχή είπα. Έληξε. 6 υπέρ 21 κατά. Απορρίπτεται. 76. Άρχεται. Έληξε. 14 υπέρ 13 κατά εγκρίνεται 77 αρχή έληξε 27 ομόφωνα υπέρ εγκρίνεται 78 άρχεται έληξε 6 υπέρ 21 κατά απορρίπτεται 79 άρχεται 26 υπέρ να εγκρίνεται. 80 υπέρ. Έλξε. 25 υπέρ μία αποχή εγκρίνεται. 81 άρχεται. Έλξε. 26 υπέρ εγκρίνεται. 82 έρχεται. 6 υπέρ 13 κατά 8 αποχές απορρίπτεται. 83 έρχεται Έλξε. 14 υπέρ, 13 κατά εγκρίνεται. 84 και τελευταία αρχίζει η ψηφοφορία. Ε, έληξε. 13 υπέρ, 12 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Τώρα το σύνολο, το σύνολο, σύνολο, έληξε. 20 υπέρ 7 κατά. Εγκρίνεται το έγγραφο εργασίας. Τους ευχαριστώ όλους. With this vote, the meeting ends. Thank you.